Right, welcome everybody. it's loud. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ε, έχει μεγάλο θόρυβο και πολύ ζέστη. Δεν ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι τεχνική. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο της ημερήσιας διάταξης 10. Τροποποίηση της οδηγίας 2006-112-6 ε, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Ο David Κάσα είναι ο υπεύθυνος αλλά σήμερα θα αντικατασταθεί. Δυστυχώς ε, υπάρχει συνένεση προς αυτό και γι' αυτό όλοι βιάστηκαν να έρθουν. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Σάρων. Όπως είπατε, ο κύριος Κάσα αυτή τη στιγμή ε, δεν μπορεί να έρθει και ζητήσε να τον αντικαταστήσω. Θα διαβάσω λοιπόν αυτό που ετοίμασε. Λάβαμε ένα σύνολο 22 τροπολογιών για αυτή την έκθεση. Λίγο πολύ ζήτησε να υπερψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες εκτός από μία. Επίσης, έχει διαπραγματευτεί τρεις συμβαστικές τροπολογίες. Μετά από τα όσα άκουσε για την τροπολογία 6 όσον αφορά στη δημιουργία κατοφλίου σχετικά με την ε, ε, μεγάλη απάτη αποφάσισε να αποσύρει αυτή την τροπολογία. Επίσης θέλει να πούμε ότι όλοι συμφωνούμε πως η απάτη για το ΦΠΑ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στεναρά και πρέπει να γίνει κάτι και αυτός ο μηχανισμός γρήγορης δράσης είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ο κύριο Κάσα θέλει να, ευχαριστήσει όλου του συναδέλφου για την ε, συνδρομή τους. Ωραία. Σύντομο και γλυκό. Όλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να πω ότι η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα υπηκοδομητική και αυτή τη στιγμή έχουμε ε, μια μεγάλη πλειοψηφία για την ε, πρόταση της Επιτροπής. Ο Μηχανισμός Ταχείας Δράσης είναι ένα εξαίρετο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και προς την ενίσχυση της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη της απάτης του ΦΠΑ. Μια πιο ψηφιακή μορφή συνάλλαγων επίσης ε, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες προσπάθειες ε, για πάταξη της απάτης ε, στο σύστημα. Και είναι πολύ σημαντικό για άλλη μια φορά να αντιδράσουμε ταχαίως. Η θέση μου εδώ σχετίζεται με μια σειρά κεντρικά ζητήματα που θα ήθελα να τονίσω στην πρόταση της Κομισιόν. Καταρχάς, είναι σημαντικό η Επιτροπή συστηματικά να διασφαλίζει ότι ο μηχανισμός θα διαθέτει όλες ε, τις δυνατότητες πάταξης της απάτης. Ε, η φορολογική απάτη είναι ένα εύκολο εργαλείο. Έχει... Μπορεί να παταχθεί εύκολα με διάφορα εργαλεία και είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών και των συμμετοχόντων. Είναι σημαντικό να υπάρχει ροή πληροφοριών σε όλες τις φάσεις για να μπορούμε να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Τρίτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι κατάλληλες διοικητικές, οι κατάλληλοι διοικητικοί πόροι στην Επιτροπή ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ταχαίως όπως σχεδιάζεται. Η Επιτροπή επίσης πρέπει να κάνει εκθέσεις τακτικά για το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός, αλλά και ο μηχανισμός πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη πάνε πιο γρήγορα πρέπει πολλές φορές να λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να πατάξουν την απάτη. Και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε πέντε μήνες. Αυτό που ε, λέγεται για τη μαζική απάτη, εγώ θα ήθελα η Κομισιόν να αποσύρει την πρότασή της. Είναι το 0,5% των εσόδων ενός, κρατού, ενός κράτους μέλους αυτό που προτείνει η Κομισιόν. Καλό θα ήταν να πάμε στην αρχική πρόταση και η Κομισιόν να ορίσει το μαζικός, ε, τον όρο μαζικός ε, στην απάτη του ΦΠΑ. Ελπίζουμε για θετικά αποτελέσματα βέβαια σε αυτό το σενάριο η συνεργασία μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθέτει προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ τον Ντέβιτ Κάσα για τη δουλειά που έκανε και για τον τρόπο που προχώρησε σε αυτό το θέμα. Ωραία. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει για αυτό το θέμα. Υπάρχει κάποιος στην αίθουσα που θέλει να μιλήσει για αυτό το θέμα. Θέλει να πει κάτι η Κομισιόν για να γεμίσει το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ναι, ευχαριστώ Κύριο Πρόεδρε. Καταρχάς να υπογραμμίσω ότι ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του και ε, με τον τρόπο που για τον τρόπο με τον οποίο έδωσε την ε, γνώμη του τον ε, συστηματικό τρόπο. Επίσης να πω ότι είχαμε μεγάλες δυσκολίες ε, για να εγκριθεί η πρόταση στο Συμβούλιο γιατί πολλά κράτη-μέλη δεν είναι υπέρ αυτού του μηχανισμού ταχείας αντίδρασης όταν αμφισβητεί την φορολογική τους κυριαρχία. Στον βαθμό δηλαδή που την αμφισβητεί. Όμως σε αυτό το στάδιο είμαστε αισιόδοξοι γιατί με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου θεωρούμε ότι η ζυγαριά θα κλείνει πιο θετικά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτά ήθελα να πω σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ και άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του. Ωραία, ευχαριστούμε. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πείτε εκ μέρους του Ντέιβιτ. Όχι, ωραία. Σας ευχαριστώ όλους. Οπότε τώρα έχουμε άλλο ένα τέταρτο μέχρι να έρθουν οι υπόλοιποι για την έκθεση του Γκούναρ. Δεν είναι κανείς εδώ, ούτε ο Γκούναρ, ούτε ο Ρουφ, ούτε ο Φίλιπ, ούτε η Βίκη, ούτε η Μαρίς. Μάλλον πρέπει να περιμένουμε. Εγώ εδώ είμαι πάντως. Συμφωνούμε επί των πάντων. Δεδομένου ότι η ώρα 9.30 ήταν ενδεικτική, ας τους δώσουμε ένα τεταρτάκι και οι βοηθοί να δουν που είναι οι βουλευτές μας, γιατί το χρονοδιάγραμμα είναι απλώς ενδεικτικό. Ευχαριστώ.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 Sí, pero ya está. Ah. Ya. Right, I think we have uh, captured enough shadows that we can now... Νομίζω έχουμε αρκετούς και οδησυγητές εδώ, τόσο ώστε να είμαι θα να προχωρήσουμε στο σημείο υπαρθμών 11, που είναι αυτή η έκθεση του Γκούναρ Χόκμαρκ, η οποία αφορά αυτό το ψήφισμα και επίσης την εκθέση των τροπολογιών. Πάρα πολύ μου ασχοληθεί με αυτήν την υπόθεση, οπότε παρακαλώ καθίστε και θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Γκούναρ. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές. Μέχρι στιγμής ε, η συμμετοχή τους, η συμβολή τους ε, με βοήθησε, με ενέπνευσε. Συναντηθήκαμε και συζητήσαμε πολλές φορές το σημείο αυτό. Οι τροπολογίες είναι πολύ άριθμες από όλες τις πολιτικές ομάδες και από όλους τους ευρωβουλευτές και είναι πολύ επικοδομητικές. Είμαι πολύ ικανοποιημένο από την υψηλή ποιότητα συνεισφορών. Και αυτό με καθιστά αισιόδοξο για το, την πορεία και το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία. Καταρχάς, πιστεύω ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι ότι αυτή η έκθεση είναι ακρογωνιαίος λήθος της ενίας αγοράς και πρέπει να αποτελέσει τμήμα της, των χρηματαγορών και να αποτελέσει και ευκαιρία για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό ισχύει εν μέρη. Γιατί? Γιατί όταν βλέπετε τις τροπολογίες καταλαβαίνετε πού προέρχονται αυτές οι τροπολογίες. Και το λέω χωρίς καμία ηρωνία αυτό. Αντικατοπτρίζουν αυτές οι τροπολογίες την πραγματικότητα των ιδεολογιών, των απόψεων για την οικονομία ε, και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτές οι διαφορές δεν αφορούν το σωστό ή το λάθος ή την διαφορετική πολιτική γεύση αφορούν την ευθύνη μας να εξετάσουμε και να απεικονίσουμε με σεβασμό τις διαφορές απόψεων που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό να το εξασφαλίσουμε. Και το αποτέλεσμα αυτού του νομοθετήματος να είναι ότι αντικατοπτρίζει και σέβεται όλες τις διαφορετικές απόψεις και καταστάσεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ακρογωνιαίος λήθος αυτό το νομοθέτημα, γιατί με αυτόν τον τρόπο αποκαθιστούμε τον καπιταλισμό Και κάθε θεσμικό όργανο, κάθε εταιρεία, κάθε διαχειριστής, κάθε διευθυντικός στέλεχος, κάθε μέτοχος έχει τη δική του ευθύνη και πρέπει να το αποδοθεί. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε. Ένα σημαντικό πράγμα είναι το πώς εξετάζουμε το τη διάσωση, η οποία διάσωση πρέπει να γίνεται με συμμετοχή και πληρωμή όλων των υπευθύνων. Αυτή η πληρωμή, αυτή η πληρωμή για τη διάσωση είναι σημαντική. Και επίσης το νομοθέτημα θα πρέπει να σου λέει πού υπάρχει, ποιο είναι το σημείο σύγκλησης. Οι επενδύσεις και πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όταν πτωχεύει μια εταιρεία, αυτοί οι οποίοι έχουν επενδύσει κινδυνεύουν να χάσουν τα λεφτά τους, φυσικά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Κι όμως αυτό είναι σημαντικό, γιατί ε, με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές πρέπει γνωρίζουν τις, ε, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Και αυτό είναι σημαντικό ε, να υπάρχει αυτή η διαφάνεια στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και τελικά είναι σημαντικό να έχουμε μια απόφαση για αυτή την ιδέα, ότι πληρώνω για τη διάσωση, ότι ο καθένας συμμετέχει για τη διάσωση. Οι, οι επενδύσεις ε, για τις τράπεζες θα πρέπει να απλωθούν σε μια πλειάδα συμμετεχόντων. Ε, και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν του, τα ρίσκα, τους κινδύνους. Επίσης, Είπαμε πολλές φορές ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι δεν τη γλιτώνει κανένας εύκολα με τα λεφτά των φορολογούμενων μόνο. Καμία τράπεζα, κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ ευρεία συνένεση μεταξύ ημών, συναδέλφων και σκιωδών εισηγητών. Και αν τελικά θέλουμε να υπάρχει ουσιαστική σταθερότητα σε τραπεζικές κρίσεις, όταν δέχεται μια συστημική κρίση, πρέπει να έχουμε και την δυνατότητα της δημόσιας παρέμβασης με κάποιο τρόπο. Να μην είναι αυτό το πρώτο βήμα, να μην είναι αυτή η εύκολη λύση βέβαια, αλλά να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα εξασφάλισης του συνολικού α, συστήματος. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια πλειάδα εργαλείων πριν φτάσουμε εκεί αλλά να έχουμε και την ε, δυνατότητα να προσαρμοστούμε. Γιατί όταν μια τραπεζική κρίση ξεσπάσει, ποτέ δεν είναι όπως την έχετε προβλέψει. Πάντα είναι διαφορετική. Η φύση της κρίσης ακριβώς αυτή είναι, ότι σας εκπλήσει. Μας εκπλήσει. Και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την ευελιξία. Μία σκέψη που έκανα για τις τροπολογίες που προήλθαν από διάφορους συναδέλφους είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για το, το σχεδιασμό μας, για το πώς θα πρέπει να επιληθούν τα πράγματα, γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να υπάρχει ευελιξία για αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση να ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν την κρίση, την ανάκαμψη και την εξυγίανση. Αυτή είναι μια ευθύνη που έχουμε συνολικά. Παρότι βέβαια κάποιες λεπτομέρειες θα πρέπει να υπάρχουν, πάντα, πάντα υπάρχει κίνδυνος να δημιουργήσουν μεγάλο βαθμό ακαμψίας και να υποσκάψουν την δυνατότητα που έχουν όσοι παίρνουν τις αποφάσεις, να πάρουν τις σωστέ αποφάσεις και έγκαιρα μάλιστα. Όπω ξέρουν οι συναδέλφοι έχουμε περίπου 1.700 τροπολογίες από όλε τι πολιτικές ομάδες και πολύ λίγες τροπολογίες είναι αντιφατικές. Απλώς ε, έχουν πολλές αποχρώσεις για το πώς μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δυσκολεύομαι μάλιστα γιατί <laughs> συμφωνώ με όλες τις ιδέες. Αυτό είναι και καλό γιατί έτσι ξέρουμε τις λύσεις. Αλλά γιατί τα λέω όλα αυτά, για να σας πω ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να επιληθεί ένα πρόβλημα. Μερικοί από αυτούς τους τρόπους μάλλον είναι πολύ καλοί και κάποιοι άλλοι ακόμα καλύτεροι. Αυτό περιπλέκει τα πράγματα. Γιατί είναι εύκολο να επιλέξουμε ανάμεσα σε μια καλή και σε μια κακή εναλλακτική λύση. Αλλά όταν έχει δύο καλέ εναλλακτικέ λύσει, το πράγμα γίνεται πιο δύσκολο και πρέπει να σκεφτεί περισσότερο. Από την άλλη, βέβαια, ε, υπάρχει και περιθώριο για πιο επικοδομητικούς συμβιβασμού και συζητήσει. Να σταθώ σε κάποια από τα θέματα που τονίζουν ε, οι τροπολογίε, Το πεδίο εφαρμογή καταρχάς. Πολλέ ε, τροπολογίε ζητούν εξαιρέσει. Λένε ότι ορισμένε εμπορικέ τράπεζες θα πρέπει να εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Γιατί ορισμένες κατηγορίες τραπεζών δεν θέτουν συστημικό κίνδυνο. Και τότε και θα ήταν δυσανάλογο να, βαραίνουν, να βαρύνουμε και με αυτές ε, το νομοθέτημα αυτό. Εγώ πιστεύω βέβαια ότι δεν πρέπει να εξαιρεθεί καμία τράπεζα αλλά και είναι σημαντικό οι αρχές να μην σπαταλούν την ενέργειά του για τράπεζες που δεν είναι σημαντικές, που δεν θέτουν δηλαδή ζητήματα συστημικού κινδύνου, που δεν αποτελούν συστημικό κίνδυνο οι ίδιες. Θα πρέπει τελικά να φτιάξουμε κάποιε εξαιρέσει, να εξαιρέσουμε, να βγάλουμε εκτό του πεδίου εφαρμογή κάποιε τράπεζε που διαφέρουν ακριβώ. Ακριβώ υπ' αυτή την έννοια από το συνήθι, τη συνήθι τράπεζα και το τραπεζικό τομέα. Επίση, ε, πώ θα υποδειχθεί η αρχή ε, εξυγίαση. Αυτό μιλάνε γι' αυτό πολλέ ε, τροπολογίε. Θα είναι μια μεγάλη τέτοια αρχή ή θα έχουμε την εποπτική αρχή και η, εποπτική, και η αρχή εξυγίαση θα εντάσσεται σε αυτήν. Το σημείο φετηρία μου είναι ότι καλό είναι να πούμε ότι διορίζουμε μία αρχή εξυγίανσης. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε και την κρίσιμη μάζα και τη γνώση και την, την αρμοδιότητα για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά να εξασφαλίσουμε και την διαίρεση, το διαχωρισμό ανάμεσα στην εποπτεία και στην εξυγίανση. Γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε να έχουμε σύγκρουση συμφερόντων. Και κινδυνεύουμε οι αποφάσεις να επηρεαστούν με λάθος τρόπο είτε από την αρχή εποπτείας, η οποία θα είναι πολύ μαλακή για τις τράπεζες κατά την εξυγίανση ή αντίστροφα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης, η τάση είναι οι βουλευτέ να λένε ότι όταν υπάρχει ένα ίδρυμα ή μια τράπεζα που έχει σημαντική, ε, σημαντική θέση σε ένα κρατός θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό σχέδιο και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από την αρχή. Είναι σημαντικό αυτό. Το δικό μου σημείο φετηρίας είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν ευθύνη για την αντιμετώπιση των πραγμάτων. Έχουν μετόχους, έτσι. Τι χώρε Ορισμένες χώρες υποδοχής τραπεζών αισθάνονται ανασφάλεια για τις ε, θυγατρικές της, ε, στην επικράτειά τους. και λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδικό σχέδιο εξυγίανσης και ανάκαμψης για σημαντικές τράπεζες στη χώρα τους. Πότε ξεκινάει η έγκαιρη παρέμβαση. Τι τη δρομολογεί. Η... Το σημείο φετηρίας για τη ρευστότητα είναι πολύ αφαίρετο. Και η πρότασή μου στο σχέδιο έκθεσής μου είναι να μην βάλουμε τη ρευστότητα σημείο αφετηρίας πολλοί συνάδελφοι έβαλαν αυτό το θέμα, ότι η ρευστότητα, το θέμα της ρευστότητας θα πρέπει να είναι ε, ένα στοιχείο που δρομολογεί την όλη διαδικασία. Ας προχωρήσουμε και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάποιο συμβιβασμό εκεί. Πρέπει όμως να μην είμαστε αφαίρετοι. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα πράγματα και να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του δικαίου για διάφορους λόγους. Καταρχήν, και για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, αλλά και γιατί όταν υπάρχει μια κρίση θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες για το πότε δρούμε και πότε δεν δρούμε. Φοβόμαστε και ανησυχούμε για το γεγονός ότι αυτές οι εξουσίες για τις οποίες νομοθετούμε μπορούν να τύχουν κατάχρησης για διαφορετικού λόγους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εκεί στο μυαλό μας η ασφάλεια δικαίου. Πιστεύω ότι η ρευστότητα δεν θα πρέπει να ξεκινά να δρομολογεί τη διαδικασία, αλλά είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Ε, γιατί από πίσω υπάρχει η ανάγκη για ασφάλεια δικαίου. Τώρα, για το ποιος πληρώνει για τη διάσωση. Το συζητήσαμε πολύ ε, με τους κοιόδης συζητητές και κάναμε ενδιαφέρουσες ε, συζητήσεις, ακούστηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες γι' αυτό. Ορισμένοι είπαν ότι υπάρχει ένα ειδικό τμήμα για τη χρηματοδότηση της τράπεζας που πάει για τη διάσωση και οι υπόλοιπες επενδύσεις δεν χρησιμεύουν για αυτή τη χρηματοδότηση της διάσωσης. Η χρηματοδότηση από τις τράπεζες τις ίδιες της διάσωσής τους είναι καλό πράγμα. Οι επενδυτές σε μια τράπεζα είναι ε, μια μεγάλη βεντάλια, μεγάλη πλιάδα. Πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο σύστημα που να καλύπτει λίγο πολύ όλη τη χρηματοδότηση της τράπεζας. Αν από την άλλη όμως όλα τα κεφάλαια πάνε για τη διάσωση, τελικά μπορεί να μην υπάρξει διάσωση, χρηματοδότηση, πραγματική χρηματοδότηση για τη διάσωση. Ο συμβασμός θα ήταν να έχουμε μια ιεράρχηση των κεφαλαίων της τράπεζας και να πούμε κάποια από τα βήματα όταν προχωρούμε προς τα κάτω στη σκάλα, κάποια κεφάλαια ας πούμε πηγαίνουν για την χρηματοδότησή της για τη διάσωση της χρηματοδότησης, δηλαδή της διάσωσης. Και επιλέγουμε το επίπεδο δράσης και απόφασης. Δεν λέμε ότι αυτά τα λεφτά πάνε για τη διάσωση. Απλώς λέμε, ιεραρχούμε τα πράγματα και λέμε, να το κεφάλαιο, τι πηγαίνει για την ε, διάσωση. Υπάρχουν βέβαια ε, ιδέες ότι όλο το κεφάλαιο της τράπεζας πηγαίνει για τη διάσωση. Με εξαίρεση το θέμα των α, κάποιων χρεών συγκεκριμένης διάρκειας. Ας πούμε, η διάρκεια μέχρι έξι μήνες, ας πούμε, μπορεί να εξαιρεθεί, χρέη μέχρι έξι μήνες μπορεί να εξαιρεθούν, ούτως ώστε να μην υπάρξει αστάθεια στην αγορά. Επίσης υπάρχει ευρεία συνένεση ότι θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους κανόνες, ούτως ώστε να μην τη γλιτώνει η τράπεζα εύκολα. Και βεβαίως, οπωσδήποτε, και οι μέτοχοι θα πρέπει να πληρώνουν αυτό που οφείλουν να πληρώνουν πριν τη δημόσια παρέμβαση. Επίσης, οι αρχές στη χώρα υποδοχής πρέπει να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες. Ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα είναι η χρηματοδότηση του Ταμείου Εξυγίανσης. Ε, το σημείο Φετηρία είναι ότι πρέπει να έχουμε μια αρχική χρηματοδότηση. Αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια ευελιξία για κράτη-μέλη που έχουν άλλη παράδοση, που έχουν άλλους τρόπους να προχωρούν. Θα πρέπει να έχουμε τα βασικά κριτήρια. Ο, ειλικρινά σας λέω, δεν ξέρω πώς μπορούμε να έχουμε συμβιβασμό για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με τους κοιόδης συζητητέ και με τους υπόλοιπου ευρωβουλευτές βέβαια. Θα σταματήσω εδώ και θα δώσω το λόγο στου συναδέλφους. Αλλά ακόμα μια φορά θέλω να σας πω ότι είμαι πραγματικά ευγνώμων για τη συνεργασία που είχαμε και με μεγάλη χαρά θα περιμένω να ανταλλάξουμε απόψει. Πιστεύω, Πρόεδρε, ότι είμαστε σε μια φάση όπου θα πετύχουμε καλούς συμβιβασμούς. Πιστεύω ότι είναι μια έκθεση υψηλή ποιότητα. Η όλη διαδικασία είναι πολύ ποιοτική και χαίρομαι που είμαι τμήμα αυτής της διαδικασίας. Λύσα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω αγγλικά γιατί όλοι είμαστε λίγο κουρασμένοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Γκούναρ για όλη τη δουλειά που έκανε για την υπομονή του, την στάση του, γιατί νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση στην ομάδα. Λίγο πολύ συμφωνώ μαζί του όταν λέει ότι κανείς δεν έχει πιστεί πως η αλήθεια βρίσκεται στη δική του πρόταση, αλλά όλοι προσπαθούμε να βρούμε κάτι που να λειτουργεί και να πετυχαίνει τους στόχους. Έχω επίσης ε, την τάση να συμφωνήσω με τον Γκούνερ όταν λέει ότι από αυτό θα βγάλουμε μια σειρά καλών συμβιβασμών. Θα προσπαθήσω να αντιδράσω στα διάφορα σημεία που ο κύριος Χόκμαρκ παρουσίασε για την κάλυψη συμφωνώ ότι κάποιες τράπεζες πρέπει να έχουν έναν πιο χαλαρό έλεγχο και ένα χαλαρό επίπεδο απαιτήσεων. Γι' αυτό θα προτιμούσα ένα ευρύτερο πεδίο σε αυτήν την νομοθεσία. Ιδάλλως θα αρχίσουμε να βάζουμε τις διάφορες προϋποθέσεις και στο τέλος ε, θα έχουμε μια αντιγραφή αυτού που τελικά εμείς προσπαθούμε να ελέγξουμε. όπου τελικά οι πιο επικίνδυνες τράπεζες θα θεωρούνται οι πιο ασφαλείς γιατί θα εποπτεύονται παγκοσμίω συνολικά μάλλον και οι άλλες όχι. Αυτό προσβάλλει την κοινή λογική. Και τελικά ε, το περιθώριο χειρισμών που έχουν ε, οι εθνικές αρχές ε, για να μην ζητούν δυσανάλογες πληροφορίες όταν δεν χρειάζονται, να μην ασκούν πίεση στις τράπεζες, η δυνατότητα να παρεμβαίνουν και να ζητούν επιπλέον απαιτήσει αν χρειάζονται, αυτό είναι κάτι που θα διακυβευτεί. Έτσι λοιπόν, αυτές οι ασφαλείς τράπεζες ε, που ασχολούνται με καταθέσεις, αν κάποια από αυτές ε, λόγω κακοδιαχείρισης ή για οποιοδήποτε λόγο έχει προβλήματα, τότε θέτει έναν πολύ σημαντικό συστημικό κίνδυνο, γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν πλέον. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, αυτό το ζήτημα αν μία από αυτές τις πολύ ασφαλείς τράπεζες έχει προβλήματα. Δεν πρέπει λοιπόν να εξαιρούνται. Χρειάζεται η εμπιστοσύνη, αλλά η εμπιστοσύνη πρέπει να βασίζεται και στη γνώση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν λειτουργεί η σκέψη μου. Ακόμα και σε χώρες που έχουμε διαφορετικές οντότητες που τελικά ε, μπλέκονται στο ε, σχέδιο ανάκαμψης ε, και εξυγίανσης, κάπου χρειάζεται να υπάρχει ένας ηγέτης, μια οντότητα που θα είναι υπεύθυνη, γιατί ακόμα και στις τράπεζες που είναι διασυνοριακές, δεν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ομιλητής εκ μέρους τους. Για τον διαχωρισμό μεταξύ της εποπτείας και της ε, εξυγίανσης να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διαφορετικές οντότητες διαφορετικ... ή αν είναι η ίδια η οντότητα να υπάρχουν ε, να υπάρχει διαχωρισμός των ευθυνών και της λήψης αποφάσεων. Πρέπει να έχουμε εγγυημένους ε, μηχανισμούς εταιρική συνεργασίας ε, για να δούμε ποιος είναι ο βαθμός δίδυσης που έχουν στην εποπτεία. Γιατί μπορεί αυτό να παγιδεύσει το αποτέλεσμα της εξυγίανσης. Και ως προς την εξυγίανση είναι καλό να γνωρίζουμε τι τελικά αναγκάστηκε να κάνει ο οργανισμός υπό την εποπτεία του εποπτεύοντα οργανισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που είναι ποσοτικοί και ποιοτικοί και που οδηγούν ε, έναν τραπεζικό οργανισμό σε προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ισορροπία. Θα πρέπει να συζητήσουμε για άλλη μια φορά την πρόταση δημιουργίας ε, ενός ε, προστατευτικού τείχους. Αυτό που είπαν οι πράσινοι δηλαδή στις ε, τροπολογίες τους. Όλες οι επαπτικές αρχές να μπορούν να εξετάζουν μια σειρά δικτών οι οποίοι θα είναι ένας πιο ισορροπημένος και ξεκάθαρος τρόπος για να εξετάζεται η υγεία ενός οργανισμού. Αυτό φυσικά δεν θα υποκαθιστά αυτά επί των οποίων έχουμε ήδη συμφωνήσει. Απλώς θα αυξάνεται τις πληροφορίες και θα δίνει σε όλους την ίδια εικόνα προς εξέταση και ειδικότερα για τα διασυναριακούς οργανισμούς θα διευκολύνει τη συζήτηση για την υγεία. Για το Μπέιλιν τα εργαλεία διάσωσης με ίδια μέσα, επίσης συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Χόκμακ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το εργαλείο να είναι ευρύ, αλλά και πολύ ξεκάθαρο σε επίπεδο ιεραρχίας. Και θα προτιμούσα να πάμε στα... στην κατεύθυνση της πρότασης Λικάνεν με λίγες εξαιρέσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται η βραχυπρόθεσμη αγορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζών. Θα πρέπει να δούμε αν θα είναι τέσσερις μήνες, πέντε μήνες ή αν θα είναι κάτι σταδιακό. Είναι σημαντικό όμως να αρέει η ρευστότητα. Θα εξαιρούσα επίσης τη χρήση του ΣΕΚ, του Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων, γιατί είναι πολύ σημαντικό να επανέλθει η εμπιστοσύνη στις τράπεζες και είναι σημαντικό να εξετάσουμε όχι μόνο τις ευαισθησίες των ε, κρατών μελών, αλλά ε, και να γνωρίζουμε γιατί γίνεται αυτή η νομοθεσία. Όταν πάει κάτι στραβά, θα πρέπει να υπάρχει και η εμπιστοσύνη στις τράπεζες είναι κάτι που πρέπει να βασίζεται στην νομοθεσία. Για τη δημόσια παρέμβαση θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι τελευταία-τελευταία λύση και η έσχατη λύση και τελικά να είναι η νομοθεσία αυτή που θα ρυθμίζει. Αν δεν υπάρχει πλέον εναλλακτική και η μόνη λύση είναι η προσωρινή δημόσια ιδιοκτησία, εντάξει. Αλλά γενικά θα πρέπει να είναι η άσχατη λύση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν καταφέρουμε να βγάλουμε τους φορολογούμενους τουλάχιστον από την πρώτη φάση. Πώς τώρα ήταν παράδοση δυστυχώς για να είναι σοβαρή δουλειά που κάνουμε πρέπει να υπάρχει αυτός ο φράχτης της εξυγίανσης. Διάφορες χώρες έχουν εργαστεί πάνω σε αυτά τα ταμεία εξυγίανσης. Δεν πρέπει να βασίζονται στις καταθέσεις, γιατί αυτή είναι η ασφαλής πλευρά της ιστορίας. Η πρότασή μας είναι η συμβολή της κάθε τράπεζας να βασίζεται στην αντίληψη κινδύνου που εισάγει στο σύστημα αυτή η τράπεζα. Θα πρέπει να δούμε ε, ποιος ε, θα είναι ο τρόπος εκπροσώπησης, ε, δηλαδή θα είναι το παθητικό της τράπεζας. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα γίνεται σταδιακά, αλλά γενικά θα πρέπει να είναι κάτι που θα περιλαμβάνεται σε ένα κοινό ταμείο εξυγένσης όταν ο χρόνος το επιτρέψει. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ελέγξουμε την πολυμορφία με τέτοιο τρόπο ώστε σε ένα ύστερο στάδιο όταν προχωρήσουμε και όταν θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξυγένσης που θα χρηματοδοτείται από τις τράπεζες να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε το ε, σύστημα και να είμαστε προετοιμασμένοι εκ των προτέρων έτσι ώστε να σπάσουμε τα, τη σχέση μεταξύ των κρατών και των τραπεζών και να μην βασίζονται πλέον οι τράπεζες ε, στα χρήματα των φορολογούμενων σε περίπτωση κακοδιαχείρισης και προβλημάτων της δικής τους ε, δραστηριότητας. Είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή που θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τον κύριο Χόκμαρ και όλους τους κοιόδης ε, για το θετικό πνεύμα σε αυτήν την ομάδα εργασίας επί της ε, παρούσας νομοθεσίας. Ευχαριστούμε την Πρόεδρα. Βολφ Κλίντς για το ΕΛΔ. Πάμε σε ευχαριστώ. Συμφωνώ με αυτά που είπε πριν από λίγο η Ελίσσα. Χάρη στον Κούναρ μπορέσαμε επικοδομητικά να δουλέψουν στην ομάδα, στις διμερείς ε, συναντήσεις, στις σωματικές συναντήσεις, ε, όλα καλά μέχρι τώρα. Τώρα όσον αφορά τα διάφορα επιμέρους ζητήματα, έχω να σας πω τα εξή. Για τις αρχές ε, της ε, επίλυσης των διαφορών θα πρέπει να υπάρχει μια αναχώρα κοντά ή στα πλαίσια της υποπτικής αρχής. Να μπορεί να υπάρχει δηλαδή στενό διάλογος. Δεν υπάρχει τεχνογνωσία από πλευρά των εποπτικών αρχών. Άρα θα πρέπει να είναι κοντά. Άρα να υπάρχει ένας αυτόνομος οργανισμός που αν όχι να συστεγάζεται, να βρίσκεται κοντά στο νοσηλευτικό οργανισμό. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, το εύρο αυτή τη ρύθμιση, ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδου τέτοια επιστοτικά ιδρύματα, τα οποία να έχουν ε, κυβερνητικέ εγγυήσει και άρα είναι ασφαλή. Επομένω, δεν χρειάζεται να υπόσχονται σε αυτή τη ρύθμιση. Και το ίδιο αφορά και αυτά τα πιστοτικά ιδρύματα, η κεντρική αντισυμβαλόμενη. Και να δούμε πώς θα δημορφωθεί η πρόταση. Όσον αφορά τώρα την ε, προπαρασκευή, για το, το, τα πλάνα για την ε, ανόρθωση, θα πρέπει... Γκούναρ, είπες ότι ε, προβλέπεται, αλλά μόνο για εξαιρετικές περιστάσεις. Είναι σημαντικό. Ας το αποφασίσουν οι αρχές σε συνεργασία με την τράπεζα. Τι ρυθμίση θέλουν. Πάντως, νομίζω ότι θέλουμε να καλύπτεται όμιλος και οι θηγατρικές. Για την ρευστότητα τώρα σε ποιο σημείο ενεργοποιείται θα πρέπει κάθε φορά που σταματά η ρευστότητα θα πρέπει να έχουμε μια, ε, μια, ένα περιθώριο ενεργοποίησης γιατί αυτό ίσως εν δυνάμει βάζει την, την τράπεζα σε κίνδυνο άρα τώρα οι πόροι για την ανόρθωση τι ταμείο θα υπάρχει. Ένα για τις καταθέσεις, ένα για την τράπεζα ή, εν, ή ενιαίο ταμείο. Η παράδοση έρχεται σε αντίθεση με την ε, ιστορία. Ανάλογα με το κατωσμένος που εξετάζουμε, γιατί το σαφές είναι ότι όπως και να συγκροτηθεί αυτό το ταμείο, για μεγάλο διάστημα στο μέλλον δεν θα έχουμε κανένα ταμείο. Δεν μπορεί να έχουμε κάποιο ταμείο που να μπορεί να διασώσει μια μεγάλη τράπεζα ή όλο το τραπεζικό σύστημα. Στην αρχή φάνηκε αυτό και βλέπουμε τώρα ότι όπου τυχόν υπάρχουν τέτοια ταμεία, όλα τα χρήματα χρησιμοποιούν κατά διαφορετικούς τρόπους στη Σουηδία για το χρέος, αλλού απλώς σωρεύονται τα κεφάλαια. Οπότε, εάν δεν χρησιμοποιηθεί έτσι όπως στη Σουηδία το χρήμα του Ταμείου, τότε δεν ωφελεί καθόλου. Γιατί δεν χρησιμοποιείται το, το κεφάλαιο έως ότου τυχόν χρησιμοποιηθεί για το σωστό σκοπό. Για να είναι χρήσιμο αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να είναι επαρκές ως ποσό. Να αποτελεί δηλαδή ένα χρήσιμο εργαλείο. Επομένως, το θέμα είναι κατά πόσον αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Μα διαπιστώσουμε ποιες είναι οι δυσκολίες και τα είδαμε και στη συζήτηση. Το πιο πιθανό είναι ότι τα κρατη δεν θα συμφωνήσουν να χρησιμοποιείτε αυτό το κεφάλαιο εκτός της χώρας στην οποία σώρευεται. για το βασικό κεφάλαιο είναι σαφές να γίνει αυτό και το εν τρίτον να αφορά τις, όπως είπε ο Πίτερ Σίμων τις ε, ασφάλτων καταθέσεων, την εγγύηση των καταθέσεων να καλύπτονται επίση από εκεί οι διοικητικές δαπάνες και να γίνεται αυτό το 0,25% με την εκ χρηματοδότηση. Να δούμε επομένως χρειάζονται ή όχι δύο χωριστά ταμεία. Και να δούμε κατά πόσο θα ισχύει διασυνοριακά ή όχι η χρηματοδότηση. Να δούμε και επίσης ποιες θα είναι οι εξαιρέσεις όσον αφορά τη διάσωση. Χρειάζεται κάτι να προβληθεί. Ομόλογα, καταθέσεις θα πρέπει να καλύπτονται. Να δούμε τώρα. 10% ελάχιστο ποσό για τη διάσωση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει στο νομοθέτημα αυτό να έχουμε συγκεκριμένο αριθμό. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι αρμοδιότητα της αρμόδιας αρχής. Εκείνη να καθορίσει το ελάχιστο χρέος πρέπει να έχει κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να υπαρχθεί στη ρύθμιση. Άλλωστε από χώρα σε χώρα ή και μέσα στην ίδια χώρα ποικίλει αυτή η ρύθμιση. Να δούμε τι θα προβληθεί για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Και να δούμε εάν κάποια τράπεζα ξεπερνά τη συγκεκριμένη κεφαλαιοχή απέτηση ανάλογα με το τι προβλέπεται στη σύμβαση της Βασιλείας τότε να ενεργοποιείται αυτό το 5%. Τελευταίο σημείο για την διαχείριση. Συμφωνώ με τον Παγκούνα όσο η τράπεζα είναι ακόμα ζωντανή, ακόμα σε μια δύσκολη κατάσταση. Αυτό απόκειται στους μέτοχου, τη Γενική Συνέλευση τους, για το αν θα αντικαταστήσουν ή όχι την διοίκηση. Και το αν θα υπαχθεί στη ρύθμιση αυτό βέβαια εξαρτάται από το τι θα αποφασίσει η υποπτική αρχή. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Φιλίπ Λάμπερτ για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να πω πρώτα πρώτα σε εσένα κάτι. Δεν καταλαβαίνω, Πρόεδρε, γιατί νομίζω ότι λέμε για το ίδιο θέμα τα ίδια επιχειρήματα για τέταρτη φορά εδώ στην ε, Επιτροπή. Και τα λέω σοβαρά γιατί Ξέρετε ότι δεν μας περισσεύει ο χρόνος, το ξέρετε καλύτερα από όλους εσείς Πρόεδρε. Δεν έχουμε χρόνο ούτως ώστε να λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Οπότε, το πιο το θα ήταν αυτή τη να την κάνουμε αφού φτάσουμε στη φάση των συμβαστικών τροπολογιών. Και δεν φταίει ο Γκούναρ με τόσες τροπολογίες ε, για να βρει συμβαστικές τροπολογίες αυτό είναι Ηράκλειος άθλος. Όλα όσα άκουσα σήμερα τα έχω ξανακούσει. Θα μπορούσα και εγώ να ξαναπώ τα ίδια. Για τέταρτη φορά. Γι' αυτό θα περιοριστώ σε λίγα. Να επαναλάβω λίγα πάντως νομίζω ότι είναι καλύτερα. Είναι πολύ μας ο χρόνος της Επιτροπής μας και πιστεύω πρώτον ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι πρόκειται για ένα κείμενο που αποσκοπεί το να μην πηγαίνουν το στη διάσωση τραπεζών. Δεν πρόκειται εδώ για προστασία από την συστημική κρίση. Αυτό δεν γίνεται έτσι με νόμο. Με αυτό το νομοθέτημα θέλουμε να προλάβουμε το να μας οδηγεί σε στιγμή κρίση συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επομένω. όλα αυτά πρέπει να αποτελούν την τελευταία, την τελευταία, την έσχατη λύση. Καλά, δεν θα κάνει κακό και μια αυτό το κείμενο. Αφού εμεί αποφασίζουμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τον ε, φορολογούμενο, τότε αν τα λέει θα κάνει μια τράπεζα, αυτή να πληρώνει την ύφη. και αν θέλουμε να μοιράσει περισσότερε τράπεζε, εντάξει. Αυτέ που κάνουν το λάθο να πληρώνουν. Το ίδιο ισχύει και για, την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Για όλου πληρώνουν οι κακοί οδηγοί. Το ίδιο ισχύει και για τι τράπεζε. Και έτσι θα συμμορφωθούν και οι τράπεζε. Η μία θα προσέχει την άλλη. Και έτσι θα αποκτήσει πειθαρχία ο χώρο και η αγορά. Αυτό είναι το πνεύμα των τροπολογιών που έχουμε υποβάλει. Στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι τράπεζες έχουν και για την ε, ανόρθωση και για την εξυγίανση κάποια προγράμματα, κάποια πλάνα. Πολλές όμως Πολλές φορές όμως οι τράπεζες, τα προβλήματα είναι τόσο περίπλοκα, τόσο μεγάλα που δεν σηκώνουν εξυγίανση, διάσωση. Και δεν θα πρέπει να διστάσουμε, να δώσουμε τα μέσα στις αρχές που αναλαμβάνουν εξυγίανση και διάσωση, ούτως ώστε να αναγκάζουν την τράπεζα να συμμορφωθεί με το πρόγραμμα, το σχέδιο που υπάρχει. <clears throat> Όλα αυτά. Αν θέλουμε να ωφελήσουμε τον φορολογούμενο. Εάν κάποιο σχέδιο κινδυνεύει να αποτύχει, δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και επ' αυτού έχουμε τροπολογίες. Κατά τρίτον, Όσον αφορά τα ταμεία της ε, ανόρθωσης και εξυγένσης, έχουμε προτείνει το να, υπάρχουν ε, αξιόπιστα, προχρηματοδοτηθέντα ταμεία. Καλά, έχουμε εδώ πέρα δύο προσεγγίσεις. Τελικά πληρώνει ο φορολογούμενος και κατόπιν εκείνος ανακτά τα χρήματά του, προσφέροντας κατά της τράπεζας. Το θέμα είναι βέβαια οι τράπεζες που κανείς μετά τη διάσωση μετά αυτές λογοδοτούν, δεν είναι αυτές που θα ήθελε κανείς ε, να κατηγορήσει για το, για το χρέος που Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι συμμετέχουν όλοι, οπότε ακόμα και τράπεζες που θέλουν να εξηγηθούν ε, εκείνες και αυτές να έχουν ε, συμβάλει. Τώρα όσον αφορά την εμπλοκή αυτών των προγραμμάτων, ταμείων, εγγύης καταθέσεων, να μην υπάρχει εδώ κίνδυνος, γιατί θεωρούμε η εξυγίνηση και ανόρθωση να μην κοστίζει πάρα πολύ, τόσο πολύ σε αυτό το Ταμείο Εγγύησης, περισσότερο από όσο η Γιατί έτσι στρεβλώνεται η λογική του, του κινήτρου. Κανείς δηλαδή να, μην πάει σε πτώχευση και να πάει σε, σε εξυγίανση διάσωση. Ή το αντίστροφο. Όσον αφορά την έγκαιρη παρέμβαση, η Ελίσσα Πολύ σωστά το τόνισε αυτό. Αφού, αν θέλουμε να υπάρχει μια ποικιλία ενδείξεων που να δίνουν το σήμα στην αρμόδια αρχή ότι κάτι πάει στραβά, θα πρέπει να το προβλέψουμε εάν το μόνο που έχουμε στα χέρια μας είναι το κανονιστικό κεφάλαιο, τότε είμαστε μαύρο-άσπρο. Ή τα πράγματα πάνε στραβά ή ου αλλά ίσως υπάρχει μια διάμεση φάση κάποιας δύσκολης στριμωγμένης κατάστασης, οπότε ίσως τότε είναι καλύτερα κανείς να παρέμβει και όχι πια όταν είναι αργά στο μαύρο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος ανείχνευσης του που πάει το πράγμα. Δεν λέμε ότι θα πρέπει όποιο, οποιοδήποτε τέτοιο, τέτοιο καμπανάκι κινδύνου να ενεργοποιεί την παρέμβαση. Δεν θέλουμε να γίνεται αυτό αυτόματα και από κάποιο υπολογιστή. Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια βεντάλια από διάφορους δείκτες που να χτυπάνε το καμπανάκι σαν αρχή ότι κάτι θα πρέπει να γίνει και θέλουμε επομένω κάποια μέσα έγκαιρης παρέμβασης που να δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές αρμόδιες για διάσωση και εξυγένση να παρέμβουν. Και πάντοτε η, εκ των προτέρων κοστίζει λιγότερο η διάσωση παρά εκ των υστέρων. Και σας τονίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τώρα όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την ρευστότητα. Να μην ενεργοποιείται λοιπόν κάποιος μηχανισμός αυτόματα με το που πέφτει κάποιο, κάποιο ίδρυμα, κάποια τράπεζα κάτω από το αρχικό, το προβλεφθέν συστατικό κεφάλαιο. Να έχουμε επομένω κάποιο είδους... Ε, Σημαντικό λοιπόν όλο αυτό για την ανόρθωση και την εξυγίανση. Α, ναι, να μην, είναι, να μην είναι οι δύο αρχέ μαζί. Να είναι κοντά, μην στη, κάτω από την ίδια στέγη. Θέλουμε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Θέλουμε να υπάρχει αντίδραση γρήγορη. Όταν επομένω φτάσουμε στη φάση αυτή της διάσωση, της ανόρθωσης, της εξυγίανση, τότε να μπορεί να πανεύει η υποπτική αρχή αλλά αυτοί μπορεί να θέλουν να καθυστερήσουν για να κρύψουν την ε, αποτυχία τους. Κοντά, αλλά όχι από την ίδια στέγη. Πάρα πολύ καλά. Μα τα είπε ο κύριος Κλίντ. Κλίντ, συγγνώμη. Επομένως, συμφωνώ και με αυτούς που είπαν ότι θα πρέπει να έχουμε λίγες εξαιρέσεις. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε κάποιο είδου περιοχές ασφαλείας εκτός του συστημικού κινδύνου. Εύχομαι να το λέμε, αλλά από την άλλη μεριά μπορούμε να πούμε όλοι να είναι ίσοι, όλοι να επιδέχονται σωτηρία, αλλά τότε είναι σαν να μην, σαν να μην σώζουμε κανένα. Εάν δεν είναι ξεκάθαρη η ρύθμιση, τότε τα προγράμματα διάσωση οι αρχέ, επειδή δεν θα ξέρουν ποιο θα, είναι, θα είναι το αποτέλεσμα δεν θα ενεργοποιούν το μηχανισμό διάσωση. Να έχουμε επομένω διαφορετικά επίπεδα του ποιο τμήμα από το κεφάλαιο από τα στοιχεία τέλο πάντων τα περιουσιακά τη τράπεζα θα επιδέχονται ή θα γίνεται να σωθούν. Βέβαια κάποιοι στείλουν ενεργητικό αποδίδουν περισσότερο. Ε, και φυσικά έτσι επιδέχονται περισσότερο ρίσκο. Αλλά δεν είναι κακό να ιεραρχήσουμε το τι έχει προτεραιότητα για διάσωση. Όλο αυτό θα πρέπει να γίνει με ξεκάθαρο τρόπο και έτσι λοιπόν να εξηχνιάσουμε το τι ρυθμίστα θα γίνει. Δεν είπαμε θέλουμε μια ρύθμιση για όλους. Είναι πολύτιμο πράγμα η ποικιλία στον τραπεζικό τομέα. Η νομοθεσία θα πρέπει να το λαμβάνει αυτό υπόψη, ακόμα και να το ενθαρρύνει την πολυμορφία. Να έχουν περισσότερη, όχι λιγότερη πολυμορφία. Θα πρέπει πάντως να είμαστε προσεκτικοί. είναι θέμα ποσοτικό. Εάν κανείς είναι 0,1% πάνω από το τεχνικό όριο, τότε κανείς να μπορεί να ενεργοποιεί το 5% αυτό δεν είναι λογικό, δεν είναι καλό. Να έχουμε επομένω δύο ε, φορείς που και οι δύο να παρέχουν κάποιες εγγύσεις. να τηρούν. Εγώ, ε, ίσως, χρειάζεται συνδυασμός των δύο κριτηρίων, δύο, δικτών. Για να δούμε την κατάσταση δύο τραπεζών. Πάντως, δεν θέλουμε όλοι να κάνουν τα ίδια πράγματα. Αυτό που θέλουμε είναι οι τράπεζες να είναι ασφαλείς. Αυτό είναι το κριτηριό μας, η ασφάλεια. Κάποιοι από εσάς θα πούν αυτό είναι επιβλαβές για την οικονομία. Είναι σημαντικό αλλά θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι τι έγινε πριν την κρίση κακές συμπεριφορές οδήγησαν στην κρίση με την υπερμόχλευση και ένα σωρό τράπεζες που ενήλυσαν με τρόπο που, που ήταν εκτός τόπου και χρόνου με δραστηριότητα οικονομική που δεν θα έπρεπε να γίνει. Έτσι έγινε αυτή η μόχλευση. Τα, τα είπαμε και χθε. Αυτό κάνει κακό στην οικονομία. Αλλά αν προσέξουμε, η απομόχλευση που έκαναν τα κράτη-μέλη, αυτό είναι που κρίνει τη οικονομία. οικονομίας. Και το ίδιο ισχύει όπως για τα κράτη, ισχύει και για τις τράπεζες. Θέλουμε το σύστημα να είναι πιο ανθεκτικό, πιο εύρωστο, πιο υγιές. Αν αυτό τώρα είναι βραχυπρόθεσμα επώδυνο, τι να κάνουμε. Ας υποφέρουν οι τράπεζες για τα μαρτήματά τους, όπως λένε και οι Γερμανοί. Φίλιπ, ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρος. Βέρνερ. Ναι, ναι, και εγώ θέλω κάτι να πω. Μετά. Έχει πει πολλά σωστό ο συνάδελφος Λάμπερτ. Καταρχάς είπε ότι ε, θα έκανε ένα θαύμα. Μίλησε 3,5 λεπτά και μετά, όσο συνέχιζε, είδα ότι εκτός από τους σκιώδους, σκιώδης, κανείς άλλος δεν είναι εδώ, γιατί κανείς άλλος δεν έχει την ευκαιρία να πει ούτε μια πρόταση. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστούμε, Βέρνερ. Και εγώ θα απαντούσα στα σχόλια που έκανε ο Φιλίπ. Ο εισηγητή και οι σκιώδε ε, πραγματικά παίρνουν τη μερίδα του λέοντο ε, από το χρόνο. Έχουμε 13.000. Ε, 1.300 ε, τροπολογίες. μια στιγμή, μια στιγμή. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανταλλάξουμε απόψεις επί των τροπολογιών. Όσοι έχουν ε, καταθέσει τροπολογίες πέρα από αυτές των ε, σκιωδών, θα πρέπει <coughs> να μπορούν να τις σχολιάσουν. Μέχρι στιγμής είμαι απογοητευμένη που δεν αναλύθηκαν κάποιες από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Δεν μπορούν όλα να τα λένε οι σκιώδεις μεταξύ τους μόνο. Δεν μπορούν τα υπόλοιπα να εκφεύγουν της ε, προσοχής του κοινού. Έχουμε πολλούς άλλους ομιλητές στον κατάλογο και αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος θα τον δώσω. Γιατί θέλω να ξέρω, ε, οι τροπολογίες Φέρμπερ, Μίτσας, Κλίντς, ε, Σίμον, Λάγκεν, Σουάμπ, εγώ κτλ. όλοι αυτοί έχουν απόψει. Ε, και όμω δεν έχει α, αναφερθεί καθόλου η άποψή του. Φίλιπ, δεν σου ξαναδίνω τον λόγο. Όχι, θα συνεχίσουμε. Σου λέω ότι αυτό το θέμα είναι σημαντικό και αν οι σκιώδεις δεν έχουν να πούν τίποτα καινούριο, stop, να μην μιλήσουν άλλο. Wow. Κυρία Φόρντ, θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική για το πεδίο εφαρμογής. Διαφορετικές τράπεζες αντιμετωπίζουν διαφορετικές κρίσεις. Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, αλλά θα πρέπει να είμαστε αναλογικοί ανάλογα με το μέγεθος τη Τράπεζα, δηλαδή ο αποκλεισμό που προτείνει ο κύριος Φέρμπερ, που δεν είναι σκιώδη εισηγητή για τις ε, δημόσιες τράπεζες, Αυτό δεν είναι σωστός. Γιατί μιλάει για κάποιες τράπεζες. Ας δούμε τι σημαίνει αυτό ο όρο σε κάποια Ακόμα και μια δημόσια τράπεζα μπορεί να ε, οδηγήσει σε σπατάλη για το δημόσιο χρήμα. Οι μικρές τράπεζες που πρέπει να εξαιρεθούν, λέει ο κ. Λάγκεν. Δεν συμφωνώ. Ναι, να έχουμε ένα λογικό ε, σχήμα, αλλά ξέρουμε ότι και οι μικρές τράπεζες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα. Για τη συμμετοχή του ε, ιδιωτικού τομέα στη διάσωση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη, θα πρέπει να είναι ευρύ αυτή η συμμετοχή, όσο πιο ευρία γίνεται η ανάγκη της επιμόλυσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει να έχουν οι αρχές εξηγίασης κάποια ευελιξία για να μπορούν να βγάζουν κάποιες υποχρεώσεις, ε, κάποια κεφάλαια δηλαδή. Επίσης η Ελίν που δεν είναι σκιώδης εισηγήτρια, επίσης έχει βάλει ανάλογη τροπολογία με τη Σελίσσα που είναι σκιώδης εισηγήτρια. Να έχουμε δηλαδή ε, για το θέμα της ε, επιμόλυσης μία ευελιξία. Ε, η εξαίρεση που λέει ότι οι καταθέσεις που καλύπτονται από την GS δεν μπορούν να καλύπτονται και επίσης η εξαίρεση του ενός μήνα σημαντική γιατί θέλουμε να μπορούμε να έχουμε βραχυπρόθεσμο ε, δανεισμό των τραπεζών στην Ευρώπη. Δύσκολη απόφαση αυτή. Δεν συμφωνώ με το ελάχιστο ποσό ότι θα πρέπει να βασίζεται στο συνολικό ύψος των ε, υποχρεώσεων. Ε, το κάναμε αυτό το, αυτή τη συζήτηση στη Βασιλεία. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού είναι μια ιδέα. Αυτή είναι πολύ άκαμπτη ιδέα, γιατί έχουμε διαφορετικά μοντέλα τραπεζών και θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια ευελιξία, γιατί αυτό το στοιχείο ε, οδήγησε, ήταν συστατικό της κρίσης. Πρέπει να τα γνωρίζουμε τις διαφορές. Η τροπολογία Μπίντεγκεν για την αξιολόγηση της οικονομικής επίπτωσης είναι μη ρεαλιστική σε επίπεδο σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ο Diego Φέιο χρησιμοποιεί το bail-in, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ε, ως ίστατο καταφύγιο. Εάν θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα δεν αρκεί αυτό. Συμφωνώ με την εισηγητή ότι δεν θα πρέπει να είμαστε άκαμπτοι για την απόφαση που πρέπει να ληφθεί και κάποιες από τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σενάρια για την ανάκαμψη κτλ. είναι πολύ άκαμπτα. Ε, Καλές συντροπολογίες σε Λίσσα. Επίσης, η ρήτρα για την δημοσιονομική ασφάλεια είναι σημαντική. Υπάρχουν πολλά θέματα που αφορούν το κράτος υποδοχής της τράπεζας, ε, ιδίως για τα νέα κρατή-μέλη. Άρθρο 15. Το ήξερα ότι αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα και βλέπω ο κ. Μάτρες και άλλοι έχουν ε, διαγράψει ε, πολλές από τις ε, ιδέες, δηλαδή κράτος προέλευσης, κράτος υποδοχής. Εγώ έχω κάνει προτάσεις για αυτά τα θέματα, ειδικά για τα νέα κράτη-μέλη θα είναι χρήσιμα, για τις καταθέσεις και πώς θα προστατεύσουμε τους καταθέτες. Και αυτό σημαίνει ότι προστατεύουμε τελικά τους φορολογούμενους οι οποίοι μπαίνουν και αυτοί. Είναι να βάλουμε, ε, να θεωρήσουμε τους ε, καταθέτες ως πρώτους πιστωτές. Και επομένως μειώνεται η πιθανότητα να διαγραφούν οι δικές τους επενδύσεις. Και έβαλα μια τροπολογία εδώ που λέει ότι τα συστήματα εγγύης των καταθέσεων θα πρέπει τουλάχιστον ε, να είναι στο ίδιο ύψο άλλων απαιτήσεων. Σε ορισμένες χώρες όπως η Πορτογαλία έχουν βάλει την προτίμηση των ε, καταθέσεων, πάνω πάνω τις καταθέσεις δηλαδή, είναι ε, ευαίσθητο θέμα στις, στην Πορτογαλία. Ε, ήταν θέμα και που το, που το εξέτασε και η Τρόικα. Υπάρχουν χώρες που το εξετάζουν ως εναλλακτική λύση για να συστήσουν τα προχρηματοδοτούμενα ταμεία. Συμφωνώ με αυτά που Μόρφερ για, τις, για το μέγεθος των ταμείων που πρέπει να δημιουργηθούν. Ξέρω πολύ καλά αυτά που είπε ο Μάριο Ντράγκη για τις ευαισθησίες της διασυνοριακής χρήσης των κονδυλίων των ταμείων. Εγώ το διέγραψα και βγάζω την απόφαση για την ε, χρήση των κονδυλίων των ταμείων Αυτή είναι δική, αυτό είναι στη δική μου τροπολογία, στη δική μου την, ε, τη σκέψη. Μπορεί να μην είναι σωστό, αλλά ξέρω ότι διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετική άποψη για το πώς θα ξαναπληρώσουν, θα αποπληρώσουν τα χρήματα που, κατα, που βάζουν οι φορολογιούμενοι. Παραδείγματο χάρη, ε, τα λεφτά του, που, του Ταμείου Εξυγίανσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, στη Σουηδία οι Γερμανοί έχουν άλλη προσέγγιση. Αντί να έχουμε ταμείο εγγύησης, εξυγίανσης που λέμε ότι παίρνει τα λεφτά, παρεμβαίνει το, το Υπουργείο Οικονομικών και αποπληρώνει τα λεφτά των φορολογούμενων. Πρέπει να τα δούμε με ανοιχτό πνεύμα όλα αυτά τα θέματα για την ε, οικονομική υποστήριξη μέσα στον Όμιλο. Κάποιες μεγάλες τράπεζες που έχουν θυγατρικές ε, αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικές στη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτές οι τράπεζες ανησυχούν για το αν αυτή η διατύπωση μπορεί να υποσκάψει την δομή τους, δηλαδή ότι είναι οργανωμένες με θηγατρικές. Θα πρέπει να ακούσουμε δηλαδή το πώς οργανώνονται οι τράπεζες ε, αν έχουν θηγατρικές, ε, ποιος έχει τη δικαιοδοσία κτλ. Για το τι δρομολογεί το Μπέιλιν. Σέβομαι αυτό που λέει ο εισηγητής, ότι πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, διαφάνεια. Η συζήτηση για τις κεφαλαιακές απαιτήσει δεν είναι το ελάχιστο κεφάλαιο, ας πούμε, από το οποίο και μετά από το οποίο και κάτω μάλλον αρχίζει να έχει πρόβλημα η τράπεζα, ε, υπάρχουν και θέματα ρευστότητα κτλ. ή και μη συμμόρφωση με κάποιου κανόνε. Όλα αυτά μπορούν να δρομολογήσουν ε, το σχέδιο τη εξυγίανση. Θα σταματήσω και να μιλήσουν και άλλοι. Ευχαριστώ, Βίκη. Χαίρομαι που σχολίασε και τι υπόλοιπε τροπολογίε άλλων. Χάσαμε και 20 λεφτά, εξάλλου από τη συζήτηση. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει στις 9 και 20 όταν σταματήσαμε το προηγούμενο σημείο, αλλά χρειάστηκε να περιμένουμε. Χάσαμε 10 λεπτά περιμένοντας και άλλα 10 λεπτά γιατί δεν ήταν όλοι σκιώδεις εδώ, παρότι ήταν ο εισηγητής. Δεν είναι πειθαρχημένο το τμήμα αυτό, πειθαρχημένη η επιτροπή αυτή. Δεν έχουμε χρόνο, βέβαια αλλά δεν θέλω να περιορίσω τους άλλους ομιλητές. Να σας πω ποιοι είναι. Olli Ludvigsen, myself, anybody else for the list. άλλος που θέλει να μιλήσει. Πίτερ Σίμον άλλος. Okay, right, so... Ωραία. Δανούτα. Ευχαριστώ, Σάρον. Στις ε, τροπολογίες μου έχω επικεντρωθεί στον πιθανό κίνδυνο της κακής ισορροπίας μεταξύ των ε, αρχών υποδοχής ε, και προέλευσης. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι γνωστό και το κατανοούν όλοι. Παρ' όλα αυτά, είναι δύσκολο να βρούμε τη σωστή νομική ισορροπία μεταξύ της, των συμφερόντων ε, ε, της μίας και της άλλης δικαιοδοσίας. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και θα υπάρχουν ε, θυγατρικές που θα έχουν πολύ σημαντικό ε, ρόλο να παίξουν στην σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χώρα υποδοχής. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα το οποίο από μόνο του θα προωθεί την αστάθεια. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα κρίσιμο καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να φέρει μια σωστή ισορροπία σε αυτό το θέμα. Θεωρώ επίσης ότι το να δίνουμε μεγαλύτερο ρόλο στις αρχές υποδοχής είναι σχετικό. Ο Γκούναρ από ό,τι κατάλαβα, από είπε, είπε για το αλλαγές στην στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και είπε ότι οι εθνικές αρχές ίσως να είναι συμπληρωματικές. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τον κίνδυνο αστάθειας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αν δεν γίνει σωστή εξέβρεση ισορροπίας. Επίσης, θα έπρεπε να πούμε ότι τελικά η αρχή υποδοχής είναι αυτή που λογοδοτεί για την εξυγίανση της θηγατρικής και η χώρα προέλευσης επομίζεται το κόστος. Ελπίζω πραγματικά λοιπόν να μην χάσουμε από τα μάτια μας αυτή την ανάγκη για μια καλύτερη και ασφαλή ισορροπία στις συμβαστικές τροπολογίες. Ελπίζω να μην χαθεί δηλαδή στη διαδικασία και πραγματικά θα ήθελα να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, να είναι μια ανοιχτή διαδικασία όπου να φαίνεται πως ε, διατηρείται η σωστή ισορροπία γιατί θεωρώ ότι αυτό συμφέρει τους πάντες σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Μάρκους. Ευχαριστώ. Και εγώ θα μιλήσω όπως ε, και άλλοι συναδελφοί σύντομα. Δεν έχει να κάνει με το πώς είναι το σύστημα στη Γερμανία. Έχουμε ε, τρεις ε, δομές, ιδιωτική, δημόσια και συνεργατική. Υπάρχει και ένας μηχανισμός διάσωσης. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχαμε μια σειρά πτωχεύσεων ε, και στις τρεις αυτές ε, κατηγορίες ε, στην Γερμανία χωρίς να πρέπει να πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Οπότε υπάρχουν συστήματα σε κράτη-μέλη που λειτουργούν. Άρα έχουμε μια σειρά από κράτη-μέλη που δεν έχουν κανένα σύστημα ή σύστημα που δεν λειτουργεί. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το άλλο που πραγματικά με ανησυχεί είναι ότι στις δημόσιες τράπεζες υπάρχει μια γερμανική ιδιαιτερότητα. Είναι οι τράπεζες αυτές οι οποίες ε, πρέπει να λαμβάνουν ε, ε, μέτρα για να προωθήσουν τις ανανεώσιμες ενέργειες, την εξυγίανση ιδιωτικών κτηρίων, ε, για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι δηλαδή δημόσιες ε, τράπεζες που δεν συγκρίνονται με τα ταμιευτήρια. Πρέπει να αξιολογηθούν διαφορετικά, γιατί αν έχουμε τις ίδιες προϋποθέσεις και διατάξεις για όλες τις τράπεζες όσον αφορά τα rescue funds, θα ήταν καλή, θα τις επιβαρύνουμε με ένα κόστος ε, που δεν ε, ανήκει στο πλαίσιο λειτουργίας τους και καλό θα ήταν να μην γίνει αυτό. Βλέπω ότι αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τον εισηγητή. Μίλησε ε, συγκεκριμένα για μια σειρά τραπεζών που θα πρέπει να εξαιρεθούν ενδεχομένω και πραγματικά επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, εφαρμόζουμε τους στόχους επιτόπου ε, με το σωστό τρόπο πάντοτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Όλα Λούτβιξον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο μειονέκτημα στην πρόταση της Κομισιόν. Ε, είναι η πλευρά των εργαζομένων που το έχουμε παραδεχθεί. Οι τράπεζες έχουν ε, ένα προσωπικό που δουλεύει σε αυτές και στον πραγματικό κόσμο ε, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους ε, πραγματικά θίγονται. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν και αυτοί να κατανοούν τι συμβαίνει ώστε να λειτουργούν με επικοδομητικό τρόπο και να διασφαλίζουν ότι αν η τράπεζα έχει δυσκολίε θα τη βγάλουν από αυτή τη δύσκολη θέση. Νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ισορροπημένη θέση και ως προς τους ε, ε, αποσχολούμενους ε, να δίνουμε πληροφορίες σε αυτούς κατάλληλες και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να συμμετέχουν για να μπορούν να παρεμβαίνουν στη διαδικασία. Στη φάση εξυγίανσης και ανάκαμψης αυτό θα πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να υπάρχει η ευθύνη αυτή ε, διαβούλευσης και ενημέρωσης ε, των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν το προσωπικό να το θεωρούμε ως κομμάτι του ενεργητικού και όχι ως έναν εξωτερικό παράγοντα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ο Βέρνερ. Θα είμαι σύντομος. Έχει να κάνει αυτό με τον ε, τομέα εφαρμογή, ο συνάδελφο Νίτρα ε, είπε όλες οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, όλες οι αξί, όλες, ε, όλοι οι οργανισμοί έκδοση τίτλων να βγουν από την οδηγία. Παρόλο που δεν είμαστε τόσο έτοιμοι να λάβουμε υπόψη μας αυτό που μόλις ο συνάδελφος Φέρμπερ σχετικά με την ευθύνη. Έχουμε, ας πούμε, τις ε, τράπεζες ε, που είναι δημόσιες ε, και προωθούν διάφορες δράσεις που εξαρτώνται από το κεντρικό κράτος ή τέλος πάντων υπάγονται σε αυτό. Αν έχουμε μια οδηγία η οποία θα θέσει σε κίνδυνο το εφιστάμενο σύστημα, τότε δεν θα εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Και επειδή εδώ και χρόνια συζητούμε ε, την οργάνωση των ταμιευτηρίων και των άλλων τραπεζών, ε, πραγματικά ε, συζητήθηκε το θέμα της ευθύνης και της λειτουργίας των αρχών εποπτείας. Υπάρχουν λοιπόν λειτουργούντες μηχανισμοί οι οποίοι που εμποδίζουν να συμβεί αυτό που μόλις περιγράψατε και θα πρέπει ο εισηγητής να λάβει υπόψη του τις διάφορες εξαιρέσεις που αναφέρονται στις τροπολογίες. Ο, αυτό το είπε ο Σέρμπερ. Το δεύτερο είναι το ερώτημα εάν ε, θέλουμε έναν ε, μεγάλο μηχανισμό ανάκαμψης Στην οδηγία ε, για τα ίδια κεφάλαια, ε, τα μεγάλα πιστοτικά ιδρύματα είναι πάνω από 17 δις. Ε, μιλάμε επίσης για 30 δις. Γενικά το θέμα είναι αν θα έχουμε μια ενιαία ρύθμιση για την περιφερειακή ευθύνη. Θα υπογραμμίζεται δηλαδή η περιφερειακή ευθύνη για άλλη μια φορά. η Northern Rock, η Dexia, η Bankia, όλες αυτές είναι πολύ πιο πάνω από το 17. Και καλό θα ήταν να έχουμε μια ε, νομοθεσία για, όλους, για όλα τα είδη πιστοτικών ενδρυμάτων. Ευχαριστώ, Πίτερ Σίμαν. Να Η ΚΑΠΕ έχει 8 δις ε, νομίζω, δεν ήταν πολύ σωστό αυτό που είπες. Αυτό που έχει να κάνει με τις ε, επενδυτικέ τράπεζες πρόθεσης δράσεων, αν δούμε τις τροπολογίες θα είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε ποιες είναι τελικά οι τράπεζες ε, που θα μπουν στο σύστημα. Να μην κοιτάμε μόνο αυτές που ήδη υπάρχουν. Ας πούμε, να μην ε, πρέπει να εξηγένουμε ε, ιδρύματα που ήδη είναι υγιή ε, και να υπάρχουν μηχανισμοί που θα ελέγχουν δημόσιοι όπως και μηχανισμοί ευθύνης. Όλα αυτά δεν είναι ξεκάθαρα. Όσον αφορά το bail-in, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προηγούμενους. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ε, αντιμετωπίσουμε τους επενδυτές ε, στην ε, Πορτογόλη, ας πούμε, και σε άλλες χώρες έχουμε μια ιδιαίτερη θέση για τους επενδυτές, το depositor preference. Σε μας σε αυτή την νομοθεσία θα πρέπει να σκεφτούμε εάν δεν θέλουμε να αποδεχτούμε τη δυνατότητα το εθνικό δίκαιο να υπάρχει για τις κανονικές διαδικασίες, τακτικές διαδικασίες αφαιρεγκαιότητας ή αν θα προτιμήσουμε το συνολικό σύστημα Αυτό που ζητά το σύστημα Πραγματικά πρέπει να το επαναλάβω, αλλά χρειάζεται. Ουσιαστικά λέει ότι ε, ότι το bail δεν αρκεί έτσι ώστε το 1% να καλύπτεται. Να είναι επαρκές δηλαδή. Να το πω και με αριθμούς. Αγαπητοί συνάδελφοι, δείτε το impact assessment της ε, Κομισιόν και συζητήστε με τους συναδέλφους από την Κομισιόν. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κρίση. Έχουμε 1% στο Ταμείο και έχουμε μια κατάσταση όπου η Κομισιόν θέλει να πάρει ε, συμμετοχή από τα κράτη-μέλη ε, που θα ανέρχεται στο 3% του ΑΕΠ σε μια φάση που τα κράτη-μέλη ε, βρίσκονται σε κρίση και υπάρχει και αυτό το Ταμείο Διάσωσης. Αυτό θα ήταν καλό να το αποφύγουμε. Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να έχουμε υψηλότερο ποσοστό στο Ταμείο, ένα έκτο της του κόστους ανακεφαλαίωσης ε, της ε, τρέχουσας κρίσης, λέει η Κομισιόν. Εγώ το έβαλα στις τροπολογίες μου να καλύπτεται να εξασφαλίσεις οι επενδύσεις και να χρησιμοποιείται το ταμείο. Δηλαδή συνολικά να έχουμε 3% το οποίο θα είναι τουλάχιστον το μισό του κόστους ανακεφαλαίωσης που θα χρειαστεί για αυτή την κρίση από τις τράπεζες. Αν είμαστε σοβαροί λοιπόν ε, και θέλουμε ε, το ρίσκο να το πάρουμε από τους φορολογούμενους και να το πάμε στις τράπεζες, θα πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον το μισά από αυτά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω κι εγώ. Έχω πολλές τροπολογίες που έχω καταθέσει και θα τις εξηγήσω. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειε τώρα εδώ. Θέλω να εκφράσω κάποιε επιθυμίε στον εισηγητή. Έχω κάποια σημεία τα οποία θα ήθελα να πω γενικά. Πολλοί από εσά μιλήσατε για το πεδίο εφαρμογή του νομοθετήματό μα τι θα πρέπει να περιλάβουμε, τι θα πρέπει να αποκλείσουμε. Νομίζω ότι τα περισσότερα θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε, αλλά συμφωνώ με την ιδέα τη αναλογικότητα. Η αναλογικότητα ξεπερνά το μέγεθο τη Τράπεζα αφορά και το επιχειρηματικό μοντέλο και το είδος της ε, τράπεζας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε όλα τα ιδρύματα χωρίς να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο κίνδυνο. Αν κοιτάξετε τα σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης, και αυτά μπορούν να είναι αναλογικά ως προς το μέγεθος και τη φύση. Δηλαδή, αν είστε τμήμα ενός, ιδρύματο, ενός ε, συστήματος προστασίας ενός ιδρύματος, αυτό είναι τμήμα του σχεδίου ε, ανάκαμψης και εξυγίανσής σας. Εξηγείτε πώς λειτουργεί, γιατί υπάρχει μικρότερη έκθεση ε, λόγω αυτών των συστημάτων. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε ώστε να πιο ευρύς. Δεν συμφωνώ δηλαδή με αυτό που είπαν ορισμένοι, ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε κάποιους. Από την άλλη, δεν λέω ότι θα πρέπει όλους να τους αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο, όλες τις τράπεζες με τον ίδιο τρόπο. Όχι. Για τις προϋποθέσεις για την εξυγίανση, δεν είμαι υπέρ του να προσθέσουμε πολλές προϋποθέσεις. Εν μέρη γιατί οι χρηματοπιστωτικές κρίσεις συνήθως είναι απρόβλεπτες, δεν υπακούν σε κανόνες. Αυτό είναι πρόβλημα. Και κάποια στιγμή οι αποπτικές αρχές και οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να έχουν τα εργαλεία παρέμβασης για να αντιμετωπίσουν τη συγκεκριμένη κρίση. Αλλά είναι μια λεπτή ισορροπία. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και εμπιστοσύνη στους επενδυτές από την άλλη. Αυτό το είπε και ο Γκούνερ, δηλαδή, ότι υπάρχουν δύο καλές λύσεις εδώ. Είτε θα έχουμε μια άκαπτη παρέμβαση με συγκεκριμένες εντολές, οι επενδυτέ ξέρουν που βρίσκονται ή θα έχετε ευελιξία <clears throat> και οι αρχέ εξυγίαση μπορούν να κάνουν ό,τι ακριβώ χρειάζεται για να προστατεύσουν του φορολογούμενους. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει αυτέ τι δύο ιδέε να τις συγκεράσουμε. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το να ξεχάσουμε την ευελιξία που χρειάζονται οι αρχέ εξυγίαση. Και παράλληλα όμω χρειάζεται να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλεια δικαίου. Ακούστηκε από τον Βόλφ ότι αν έχεις περισσότερα κεφάλαια, τότε αυτό μπορεί να ληφθεί. Υπόψη σε αντιδιαστολή με τον Μπέιλιν. Ε, φυσικά, λογικό είναι αυτό. Για τις ε, προληπτικές εξουσίες, ε, απορρέει από τα προηγούμενα που είπα, ότι θέλω να υπάρχουν ισχυρές τέτοιες εξουσίες πρόληψης των κρίσεων. Και αν είναι αποτελεσματικές αυτές οι εξουσίες αναγκαστικά είναι παρεμβατικές. Θα πρέπει να βρούμε την ε, ισορροπία ανάμεσα στην παρεμβατικότητα και στην αποτελεσματικότητα. Διερωτώ με Γκούνα, αν ε, είσαι λίγο πολύ υπερβολικά υπέρ της ε, μεγάλη παρέμβαση. Και δεν θα ήθελα τελικά να φτάσουμε στην εξυγίαση, όπου η εξυγίαση εξορισμού είναι πολύ παρεμβατική. Επομένως, θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία εκεί, ε, στο επίπεδο που είπα. Συμφωνώ με την αντίθεση του να βάλουμε τα κρατικά εργαλεία στην εργαλειοθήκη, ε, το να έχουμε εργαλεία κρατικής χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης δεν είναι η καλύτερη οδός για μένα. Ε, η προτίμηση των καταθέσεων αναφέρθηκε, θα πρέπει να κρατήσουμε και εδώ την ευελιξία, δηλαδή να δίνουμε σημασία στην εμπειρία των κρατών μελών, ιδίω αν πρόκειται για κάτι που επιβλήθηκε, όπως την περίπτωση της Πορτογαλίας, ας πούμε. Νομίζω ότι έτσι καλύπτονται και τα περισσότερα από τα θέματα για την ε, τραπεζική αρχή. Έχω και διάφορες άλλες προτάσεις. Επίσης, ε, υπέβαλα και τις λεγόμενες τροπολογίες ε, του Προέδρου για τις κατεξιοδότηση πράξης, ούτως ώστε να έχουμε ένα σωστό χρονοδιάγραμμα και να μην έχει τη δυνατότητα η Κομισιόν να μας υποβάλει απίστευτα πολλές κατεξιοδότηση πράξεις λίγο πριν τις διακοπές. Ε, ξέρω ότι έχουμε κάποιες διαθεσμικές συμφωνίες που προσπαθούν να ρυθμίσουν αυτά τα θέματα, αλλά συνήθω δεν λειτουργούν. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ε, να ξέρουμε πότε υποβάλλονται οι κατεξουδότηση πράξεις. Νομίζω ότι και αυτό είναι τμήμα του εφνομοθετήν. Αυτά ήθελα να πω και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στον Κούναρ. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις σας. Θα ήθελα να σας πω ότι στην εισήγησή μου το είπα σε σχέση με ένα σωρό τροπολογίες από όλους τους συνάδελφους, από όλες τις πολιτικές πτέρυγες και επίσης να σας πω ότι βλέπετε εδώ πέρα τι σχήμα αναδύεται ανάλογα από την πολιτική σας ε, προέλευση προτείνετε τις λύσεις και τόνισα τότε ότι αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει κανείς να ειρωνεύεται γιατί αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, την αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις που θα πρέπει να τις καλύψουμε και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι θα βγει ό,τι το καλύτερο από αυτή την διαφορά. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι η λύση είναι μία και ενία. Θα πρέπει επομένω να εξασφαλίσουμε ότι θα εξαλείψουμε τα σημεία τριβής και προστριβής, αλλά όμως να ξέρουμε την αφετηρία. Ότι όταν έχουμε κάποια θεσμικά όργανα που, ε, ε, στα, στα οποία υπάρχει ένας μηχανισμός ε, λίανσης των διαφορών και με κάποιο τρόπο κατ' εξαίρεση ή αλλιώς όλοι μαζί συμβάλλουμε στο να δημιουργήσουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε τέτοιες σκέψεις μετά την συζήτηση αυτή. Για ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις ε, τροπολογίες. Τότε βλέπετε κάτι το οποίο το ξέρετε, δεν είναι καινούργιο σας. Ότι δεν είναι εύκολο μια απομονωμένη τροπολογία να την λάβει κανείς υπόψη. Πολλές φορές οι τροπολογίες δεν είναι απλώς μια απλή προσθήκη, έχουν πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Και γι' αυτό σας το τονίζω με μεγάλη μου χαρά συναντήσω τους αδέλφους που θα θέλανε να μου πούνε δύο λόγια παραπάνω. Γι' αυτό σας λέω ε, ότι από πολλούς αδέλφους υπάρχουν κάποια πάγια στοιχεία που αναδύονται. Όπως μερικά πράγματα δεν είναι θέμα κυριαρχίας των μελών. Είναι το πώς θα υπάρχει μια εξισορρόπηση δίκαιη σωστή στη ρύθμιση που θα προτείνουμε. Και το πρόβλημα είναι ότι σε κάποια κρατημέλη οι θηγατρικές είναι πάρα πολύ σημαντικές για την τραπεζική αγορά, την τραπεζικό τομέα και αυτό θα πρέπει να το υπόψη. Αλλά πάντως η βασική αφετηρία είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το group γιατί εκεί, εκεί έγκυται η μεγαλύτερη ευθύνη. Και ακριβώς την ευθύνη την έχουν οι ιδιοκτήτες και οι μέτοχοι. Και να δούμε πώς θα βρούμε, πώς η κυρία Στανίτα, την σωστή ισορροπία. Να δούμε πώς θα το πετύχουμε. Επίσης, κάτι άλλο όλοι εδώ έτσι είμαστε σαν αρχιτέκτονες, σαν σχεδιαστές, σχεδιάζουμε, χτίζουμε το μέλλον. Και όσο πιο λεπτομερής και ενδελεχής είναι η νομοθεσία, τόσο περισσότερο θα καλύψουμε τις αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν σε κάποια μέλουσα κρίση, για την οποία δεν ξέρουμε. Πού να ξέρουμε. Εξασφάλιση διευκρίνηση, ισορροπία, εξασφάλιση ότι μπορούμε να διχειριστούμε οποιαδήποτε κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας υπενθυμίζω, συνάδελφοι, επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ βασικό. Το λέω αυτό στη συνέχεια των όσων είπε πρόεδρος. Υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας τραπεζικής κρίσης και μιας άλλης. Και Να, τι είπαν στην γιατί τη είπα. Είπαν εύκολα και θα γίνει η εξυγίνηση διάσωση χωρίς παρέμβαση κρατική. Σας υπενθυμίζω όμως ότι η κυβέρνηση η Αμερικανική έριξε τόσα χρήματα ώστε δεν έχουν πέσει ποτέ στις τράπεζες. Δεν νομίζω όμως ότι έτσι θα πρέπει να ενεργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν, ε, υπάρχει δημόσια επανέβαση πολλών ειδών. Είμαστε θεροβάμονες, ας κάνουμε μια ρύθμιση γιατί όταν έρθει η πραγματική κρίση, τότε θα είναι η ανάγκη πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε ταμείο εξυγείας και διάσωσης. Μα τις οικονομίες μας τις τροφοδοτεί, τις, τις τραπεζικό σύστημα, εξορισμού επομένω. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα φροντίσουμε και από αυτή, με αυτή την έννοια την σταθερότητα. Άρα, θα πρέπει επομένω να προστατεύουμε και τον προτέρων την τράπεζα, εξασφάλιση. Αυτό σημαίνει το εργαλείο του Βερολίνου και τα άλλα εργαλεία. Να έχουμε επομένω όλα τα εργαλεία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κρίση όταν έρθει και επίση ξεκάθαρου κανόνε. Κάθε φορά που υπάρχει μια μεγάλη κρίση χρειάζεται δημόσια παρέμβαση. Εάν δεν υπάρχουν τα μέσα, τότε αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία των τραπεζών και του συστήματος. Δεν λέω τι θα, θα έχουμε ως μέρος εργαλείο σε πρώτη φάση ή σε δεύτερη φάση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό μιλούμε για τραπεζική ένωση. Στις χώρες εκείνες όπου είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας όσον αφορά τέτοιες, ε, τέτοια, τέτοια διαχείριση, ε, τότε έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, που φυσικά και αυτό αποτελεί δημόσια παρέμβαση. Γιατί και αυτός ο μηχανισμός χρηματοδοτείται από τους φορολογουμένους. Και προσέδωσε αξιοπιστία στο ευρωπαϊκό σύστημα. Να είναι διαθέσιμος ο μηχανισμός και σε πρώτο επίπεδο, σε επίπεδο κρατών μελών. Αλλά ο μηχανισμός δεν αποτελεί ιδιωτική πρωτοβουλία. Ό,τι και να πείτε. Άρα είμαστε ρελιστές για όλα αυτά. Τέλος. Κάτι τώρα για την ενεργοποίηση, ή τι συνεργοποίησεις. κατόπιν των όσων άκουσα. Μπορεί κανείς να αντιστρέψει το επιχείρημα και να πει ότι τότε επιφυλεί αυτό το να έχουμε μια, μια έτσι, βεντάλια από επιλογές. Και κατόπιν μετά να έχουμε πιο σωστέ αποφάσει πολλέ φορέ. Όσο περισσότερου δείκτες και κριτήρια έχουμε, τόσο πιο δύσκολο κανεί είναι να αποφασίσει πώ θα ενεργήσει. Όσο πιο πολλά κριτήρια, τόσο πιο εύκολο είναι κανεί να καταλήξει στο ότι δεν χρειάζεται να ενεργήσει. Τώρα φαίνονται όλα σαφή. Και άρα παίρνει κάνει σωστές αποφάσεις. Όσο πιο πολλά κριτήρια, τόσο πιο δύσκολο είναι το να καταλήξει κανείς σε μία και μακάρι τη σωστή απόφαση. Πολλά κριτήρια, πιθανή αδράνεια. Άρα, ας έχουμε τα κριτήρια, αλλά να ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να ληφθούν οι αποφάσεις την ώρα της κρίσης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αδέλφους για τη συζήτηση και εγώ περιμένω πώς και πώς να τα ξαναπούμε και διμερώς και στην Επιτροπή. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε Γκούνα. Η 21η Μαρτίου θα γίνει η ψηφοφορία, είπαμε, ή κάποιες ψηφοφορίες, οπότε έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να βγουν οι συμβαστικές τροπολογίες στην Επιτροπή μας γιατί βεβαίως θα πρέπει πριν φτάσουμε στην ψηφοφορία να είναι ξεκάθαρο πώς λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας. Και μετά θα πάμε στην ε, Ολομέλεια 1η του Ιουνίου. Καταρχήν, αν λειτουργήσει αυτό το χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Πάμε τώρα στο επόμενο ε, θέμα μας, το υπαρθμό 12, η ατζέντα για επαρκής ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις. Η είναι ο κύριος Τόμας Μαν. Παρακαλώ, σε αποχρούν την αίθουσα, να μην κάνουν θόρυβο, γιατί εδώ θα πρέπει να φωνάζει ο Τόμας. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Στην... Η ημερήσια διάταξη για υπαρκή ασφαλή και βιώσιμες συντάξεις υπάρχουν ε, ζητήματα τα οποία ε, προκύπτουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια μια λευκή βίβλο που είναι ιδιαίτερα αμφισβητούμενη και έχουμε μια καλή ευκαιρία ε, στην ΕΚΟΝ και στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ε, έχουμε την δυνατότητα με τις δικές μας αρμοδιότητες και τις διαχωρισμένες αρμοδιότητες που έχουμε Ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Έχουμε 135 τροπολογίες και θεωρώ ότι με πολλές ε, να κάνουμε κάποια πράγματα για τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα μπορώ να συμφωνήσω από το ΕΛΚ επίσης για τη 10, 18 και 23 τη συνάδελφο Κάριν ε, έχει αναφέρει και αυτή κάποια παραδείγματα για τους σοσιαλδημοκράτες έχω προβλήματα μόνο με τον συνάδελφο Γκούτες την 13 έχει καταθέσει. Ζητά από τα κράτη-μέλη να είναι να ζητεί από τα κράτη-μέλη να θωρακίσουν ε, τα συστήματά τους ενάντια των δημογραφικών εξελίξεων και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε ε, συμβιβασμό. Η 120 επίσης μιλά ε, για το προσδόκιμο ζωής ε, και την ε, ηλικία σύνταξης. Την 29, 30 και 31 συμφωνώ για την Ούλε Λούτβιχ που δεν τη βλέπω εδώ ο σκιώδη των σοσιαλδημοκρατών. Και στον πρώτο και στον τρίτο πυλώνα έχει καταθέσει κάποιες ε, τροπολογίες την 7, την 24, την 27 μπορώ να τη δεχτώ. Για το ECR, συνάδελφος Καμάλε, τον είδα να μπαίνει, ναι, στον πρώτο πυλώνα, στην 9, 15 και 22, γιατί αυτό που προβάλλει συμφωνεί με τη σκέψη μου. Φίλιπ Λάμπερτ, σε είδα, και Φίλιπ Κρούν. Πολλές τροπολογίες από εσά, ε, πολύ μεγάλες, με το μεγαλύτερο κομμάτι συμφωνώ, από το 2 στο 4 κανένα πρόβλημα, αλλά στο 19... Έχω πρόβλημα ε, λόγω της διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Επίσης, ε, ο συνάδελφος Κρουμάν έχει καταθέσει μια σειρά τροπολογιών με τις περισσότερες δεν έχω πρόβλημα, σε δύο-τρεις υπάρχει. Η ένα, στην πυλώνα 1 για το νομοθετικό κομμάτι. Με την 25 έχω πρόβλημα γιατί ρυθμίζει πάρα πολύ από τη δική μου άποψη όσον αφορά την 11 ε, και 12 της Προέδρου την υποστηρίζω, αλλά ανήκουν στους πυλώνες 2 και 3, νομίζω. Οπότε αυτό μπορούμε να το λύσουμε. Μετά στον πυλώνα 2 έχουμε τη μερίδα του Λέοντος εδώ. Για το ΕΛΚ η Ντανούτα και η Κορίν, ο Βόρτμαν Κόλ έχουν καταθέσει πολλές τροπολογίες. Συμφωνώ με όλες, μόνο με μια λεπτομέρεια θέλω να συζητήσουμε. Ε, Ζάιτ Καμάλα από το ECR, δεύτερος πυλώνας, 100% συμφωνώ και χαίρομαι πολύ. Πρόκειται ε, για μια ε, οδηγία αναθεώρησης των συντάξεων θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο θέμα και συμφωνώ. 38, 40, 49 ε, και τα λοιπά. Για το Φίλιπ, ε, για την τροπολογία 46 έχω κάποια προβλήματα για την ρυθμιστική εναρμόνιση. Έχουμε διαφορετικές θέσεις που πρέπει να τις εξετάσουμε. Είμαι κατά μίας εναρμόνισης και μίας ρύθμισης. Είχαμε ήδη ε, στην πράξη εμπειρία εδώ στις Βρυξέλλες ε, με τις ε, συντάξεις θέλουμε μία ρύθμιση η οποία να μπορεί να καλυφθεί οικονομικά με λογικό τρόπο και αν χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις, ε, ε, ίσως ε, να χρειάζονται κάποιες εταιρείες συντάξεων οι οποίες δεν υπάρχουν. Επίσης, θεωρώ ότι η θέση του όλα είναι πολύ σημαντική και φυσικά πρέπει να δούμε αν σε κάποιους τομείς ε, πρέπει να υπάρχουν ναι, συγκεκριμένες ρυθμίσεις και θα είναι καλό να έχουμε μια συμβαστική λύση εδώ. Για το σημείο 10 θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να έχουμε συμβιβασμό. Μετά, Φίλιπ ε, Προυν, για την 55 την αποδέχομαι πλήρως θέλει μια ελάχιστη ρύθμιση των ε, απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε πόσο αυτό θα συνάδει με την πραγματικότητα. Στην 70 δεν καταλαβαίνω ακριβώς αν είστε υπέρ ή κατά της ε, χρήσης ε, του συστήματος αυτού, της φερικιότητας. Επίση ε, θα δούμε αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δεύτερο πυλώνα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το θέμα του ολιστικού μοντέλου ε, ισολογισμού με την 86 ε, ας πούμε έχω ε, συμφωνώ και με την 101 και την 110 επίσης. Όσον αφορά τις ε, τροπολογίες από το ALDE, έχετε δώσει έμφαση στο θέμα του δεύτερου πυλώνα. Συμφωνώ με τις ε, τροπολογίες 42, 51 κτλ. Το ξέρω ότι είμαι επιγραμματικός, αλλά πρέπει να πω τα σημαντικά για τον Όλε Νούκη Επίσης, ε, είναι στην ίδια γραμμή και είναι σημαντικό και αυτό που έκαναν οι συνάδελφοι οι Γερμανοί με την 67, 65 και 82 με την ε, αναθεώρηση της οδηγίας με την οποία συμφωνώ πλήρως. Έχω κάποια προβλήματα με την Γκουέ, Τόμας Χέντελ. 47 και 42 θα ήθελα αντί για ε, σύσταση θα ήθελα να αντί για σύσταση να υπάρχει ε, οδηγία. Αυτό δυστυχώς ε, το αρνείται το Solvency 2. Και για τον τρίτο πυλώνα, για τις ε, τροπολογίες της Δανούτα και της Κορίνα από το ΕΛΚ συμφωνώ πλήρως για τις τροπολογίες του Καμάλ μέχρι την 102 μπορώ να τα υποστηρίξω ε, εκεί που ζητείτε η κατάργηση του πρώτου πυλώνα υπέρ του δεύτερου και του τρίτου εντάξει ε, δεν έχουμε διατυπώσει διαφορετικά συστήματα κατά τη γνώμη μου επίσης ε, στο 33 για την εξέταση των κωδικών συμπεριφοράς Καταλαβαίνω το θέμα της ρύθμισης, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο και ρεαλιστές για να συμφωνούμε όλοι. Άρα πρέπει λίγο να το εξετάσουμε. Όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα και την ΚΟΕ, συμφωνώ με τις τροπολογίες ε, του Τόμας Χέντελ. Από την 114 έως 117 και ε, με την 131, αλλά οι κώδικες συμπεριφοράς είναι τελείως ε, μακριά από αυτό που θέλουμε, στην τροπολογία 125, για παράδειγμα. Επίσης, ε, στις διάφορες ομάδες και στους σκιώδεις ε, υπάρχει το θέμα της άρνησης του Solvency 2. Αν περάσει, αν υπάρχει πλειοψηφία, θα είναι μια, ένα θετικό μήνυμα από την Επιτροπή μας γιατί θα πρέπει να είμαστε ε, ρεαλιστές ως προς τις ε, ε, εταιρικέ συντάξεις. Για το ECR και την GUE υπάρχουν κάποια σημεία στο δεύτερο πυλώνα που πρέπει να εξετάσουμε. Έχουμε τις αποκλειστικές αρμοδιότητες στην τομέα της φεργιότητας 2 που αμφισβητούνται, θα πρέπει σε συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης να συζητήσουμε το θέμα. Τους βλέπω εδώ. Θα ήθελα λοιπόν τις επόμενες ημέρες να έχουμε μια κοινή συμβαστική λύση μαζί με τους σκιώδεις, να υπάρχει κοινή γραμμή. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές που έχουμε ακόμα, αλλά με αυτά, κυρία Πρόεδρε, ε, πραγματικά χαίρομαι ε, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Εκτός από τους Σκιώδης, δεν ξέρω ποιος άλλος θέλει το λόγο. Η Σιλβή. Άλλος κανείς. Κανά άλλο. Αν θέλει κάποιος το λόγο να μας το πει, γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Από τους σοσιαλιστές. Όλοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω πέντε σημεία τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω. Είναι σημαντικό να πούμε ότι για να λύσουμε εδώ το βασικό θέμα είναι να αυξήσουμε το, πραγματικά, το πραγματικό συνταξιδοτικό όριο. Θα πρέπει να έχουμε μέτρα, θα πρέπει να βελτιώσουμε το εργασιακό περιβάλλον, ούτω ώστε ε, να μπορούν οι άνθρωποι να δουλεύουν μέχρι την τόριο υποχρεωτική συνταξιοδότηση και να μην αναγκάζονται οι περισσότεροι να φεύγουν πριν από το όριο αυτό. Επίση, για την ποιότητα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Ποτέ δεν θα έχουμε βιώσιμες και μακροπρόθεσμες συντάξεις χωρίς να έχουμε πιο ε, ισότιμη αγορά εργασίας και προσαρμογή και συμπερίληψη στην εξίσωση των περιόδων όπου πρέπει να φύγει κανείς από την αγορά εργασία για να φροντίσει τα παιδιά του κτλ. Επίσης, οι συντάξει ηλικίας... Τι γίνεται σε περίπτωση που η εταιρεία είναι αφαιρέγγια, η εταιρεία στην οποία δουλεύουν. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους ε, εργαζόμενους για να προστατεύσουμε περισσότερο, τους προστατεύσουμε περισσότερο. Η Κομισιόν μιλάει για τις εξελίξεις των ε, υπηρεσιών ε, εποπτείας των συντάξεων. Θα πρέπει τα εθνικά συστήματα να τα διασυνδέσουμε ε, να υπάρχει μια διασύνδεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αν κάποιο δουλεύει σε διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε, α πούμε, θα πρέπει τελικά να μπορεί να ξέρει τι συνταξιδοτικά δικαιώματα έχει κατοχυρώσει. Είναι πολύ σημαντικό για την ελεύθερη κυκλοφορία στην ελεύθερη αγορά. Και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό στοιχείο της συζήτησης, που είναι το εξής. Τι θα κάνουμε με το ποσοτικό στοιχείο της εποπτείας του ταξιδιωτικού συστήματος. Πολλοί παράγοντες έχουν ε, εμπλακεί εδώ και ορισμένα στοιχεία και ορισμένα επιχειρήματα είναι πολύ απλοϊκά. Θα πρέπει να εξορροπήσουμε διάφορες ανάγκες. Από τη μία, η Κομισιόν στη Λευκή Βίβλο λέει ότι η οδηγία για τις ε, συντάξεις ηλικία θα πρέπει να κατοχυρώνουν ισοτιμία να είναι μάλλον σε ισοτιμία με το Φερεγγιότητα 2. Και τα ποσοτικά στοιχεία του Φερεγγιότητα 2 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχετικό νομοθέτημα για τις συντάξεις. Στη δική μου τροπολογία κάνω μια, μια διάκριση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες και στις υπόλοιπες εταιρείες. Μια άμεση εφαρμογή του Φερεγγιότητα 2 στη δική μας περίπτωση είναι προβληματική για τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι ένα βάρος το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε. Πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές και να βρούμε μια καλύτερη ισορροπία προετοιμάζοντας την εποπτεία των συνταξιδοτικών συστημάτων. Θα πρέπει να δούμε τις ποσοτικές προϋποθέσεις που διευκολύνουν τη λειτουργία των συνταξιωτικών συστημάτων. Η προσέγγιση με το ολιστικό, του μοντέλου ε, του ολιστικού ισολογισμού εξασφαλίζει την ασφάλεια ε, του συνταξιωτικού συστήματος και αυτή η προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική από την προσέγγιση του φερεγγιότητα 2, του κειμένου αυτού. πρέπει να κάνουμε μια μελέτη αντικτύπου για τα ποσοτικά στοιχεία. Οι ποσοτικές απαιτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αν δεν έχουμε στοιχεία για να βασίσουμε σε αυτά το νομοθέτημά μας. Πολλοί εργαζόμενοι ζημιώνονται όταν τα συνταξιδοτικά τους, ας πούμε, ταμεία ε, πλήττονται από κρίσεις. Όπως συνέβη το 2008 και 2009, δεν θέλουμε κάτι να επαναληφθεί, να την πληρώσουν τα συνταξιδοτικά ταμεία. Είναι σημαντικό τα συστήματα για τα συνταξιδοτικά ταμεία να κινούνται μέσα σε ένα πλαίσιο, να τυχάνουν τέτοιας διαχείρισης που όταν έχουμε χαμηλές αποδόσεις στις ε, χρηματαγορές, παρόλα αυτά τα ταμεία αυτά να μπορούν να επιβιώνουν. Και τα ταμεία αυτά να μπορούν να παίζουν το δικό τους ρόλο στην ε, σταθερότητα της ε, οικονομίας και των χρηματαγορών. Γιατί είναι πυλώνας του όλου συστήματος αυτά τα ταμεία, τα συνδεξιωτικά ταμεία. Και πρέπει να δούμε πώς θα τα ρυθμίζουμε αυτά τα ταμεία. Μία επικαιροποίηση της οδηγίας για τα συνδιοξιδικά ταμεία θα πρέπει να μπορέσει να δημιουργήσει μια πραγματική ενιαία αγορά που λειτουργεί απρόσκοπτα. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα σωστό, βαθμονομημένο, εύρυθμο για τα συντεξιδοτικά ταμεία. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, καλή ανάλυση των τροπολογιών που έκανε για το θαυμάσιο κείμενο το οποίο υπέβαλε και περιμένουμε να έχουμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις για την δημιουργία ε, τροπολογιών συμβιβασμού. Η Σόφη από τους φιλελεύθερους. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για τα όσα είπε για τις ε, τροπολογίες. Και εγώ περιμένω από και πώ να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε. Απλώ έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θέλω να προσέξουμε. Νομίζω ότι θέλω να πω αυτά περίπου είπε και ο προηγούμενο ε, ομιλητή, διότι στι κάτω χώρε έχουμε ένα σύστημα ε, με το οποίο δεν είναι το pay you go, είναι τα ταμεία και ε, ίσως όπως λένε το καλύτερο σύστημα στον κόσμο αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχετε τα ευάλωτα σημεία του και τα πρόσφατα χρόνια φάνηκε ότι όταν έρχεται η ώρα της κρίσης τα τα ταμεία είναι ευάλωτα και επίσης νομίζω ότι πολλές φορές εθροτυφλούμε σε σχέση με αυτούς τους κινδύνους. Ότι καμιά φορά δεν είναι καν κατανοημένοι σε αναγενές και οι μέλλοντες συνταξιούχοι, οι νεότερες γενιές έχουν πολύ μεγαλύτερη ρίσκα και τελικά δεν εκπροσωπούνται στα κέντρα τροποφάσεων, Δεν είναι οι πολιτικοί οι οποίοι ε, λαμβάνουν τις αποφάσεις. Δεν είναι η, τα, τα συνδικάτα, δεν είναι η ανώση των εργοδοτών. Τις αποφάσεις τις ε, λαμβάνουν αυτοί οι οποίοι θίγονται λιγότερο και όχι οι νεότερες γενιές που όλο για αυτές λέμε ακόμα και αν όπως είπαμε την περσμένη εβδομάδα είχαμε αυτή την ε, μελέτη ε, την Ολλανδική που έλεγε ότι ο 25 πληρώνει ακριβώς τα ίδια χρήματα σε ένα στρατιωτικό ταμείο αλλά για περισσότερα χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως θα πάρει πολύ λιγότερα από όσο ο συναδελφός του, ο οποίος είναι 20 χρόνια πιο μεγάλος. Αυτό είναι, είναι μια τεράστια δικία Και επομένω ε, θεωρώ ότι αυτές οι πτυχές δεν έχουν ε, φωτιστεί όσο θα έπρεπε ε, από τη συζήτησή μας. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε καινούργιες μορφές εργασίας, έχουμε πολλούς ε, οι οποίοι μπορεί να μετέχουν σε ένα τέτοιο ταμείο, αλλά δεν εκπροσωπούνται. Έχουμε 60, 60 εκατομμύρια οι οποίοι όμως ενθελοντικά ή επιπληρωμοί δουλεύουν εκεί και οι οποίοι όμως δεν εκπροσωπούνται. Δεν εκπροσωπούνται στα, στα ταμεία. Επομένως, ε, συμφωνώ γενικά με τον εισηγητή, αλλά κανείς εδώ πέρα από εμά δεν είπε ότι θα πρέπει ε, αυτή την πτυχή δεν, δεν έχει τονίσει. Αυτό θα πρέπει να μπει στη συζήτηση, αυτό το θέμα του κινδύνου. Το πώς θα εξασφαλίσουμε τα ταμεία να έχουν μια σταθερότητα. Και όχι μόνο όμως για αυτούς οι οποίοι τώρα είναι οι δικαιούχοι, αλλά και για τις μέλουσες γενναίες. Γιατί έχουμε επομένω ε, κάποια στοιχεία ε, τα οποία ε, όπως προβλέπει η, η συνθήκη για την αξιοπιστία 2 θα πρέπει να υπόψη. Λέμε λοιπόν τι θα γίνει, τι θα γίνει με τους μετόχους, ε, το λέμε για άλλες. Αλλά όμως η κατανομή του κινδύνου, ε, ακριβώς όπως λέμε και για τους μετόχους, θα πρέπει να αφορά και τις διάφορες επιμέρους γενναίες. Συμβολή. Και όλου. Αυτό λείπει από τη ζήτησή μα. Επομένω, αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να καταλήξουμε σε κάποιε συμβαστικέ διατάξει οι οποίε να λαμβάνουν υπόψη αυτά τα στοιχεία. Και Πάλι θεωρώ ότι έχουμε κάποιε τροπολογίε και συνεχώ λέμε για το, για αν θα ισχύσει αυτή η συνθήκη να εξούψει. Το λέμε, το ξαναλέμε. Να μην υπάρχει κανένα είδου ανεύθυνη διαχείριση γιατί την ύφη την πληρώσουν οι μελλοντικέ γενναίες. Πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε. Φίλιπ. Τόμας. Μας τα εξήγησες όσον αφορά τις τροπολογίες. Παρά τις διαφορές μας νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για τη σοφία. Αυτά γιατί γιατί συνθήκη η αξιοπιστία 2 με προβληματίζουν. Μήπως είναι λάθος ε, συνθήκη. Δεν νομίζω ότι προσφέρει ασφάλεια. Αν προσέφερε ασφάλεια, γιατί να μην ίσχυε και για τα στεξιωτικά ταμεία. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το τόσο ξεχωριστό, το ειδικό. Περίεργο μου φαίνεται εμένα που δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Φυσικά αυτό το οποίο μας λέτε είναι αφού υπάρχει ο ίδιος κίνδυνος, το ίδιο ρίσκο, ας ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Και εμείς επομένως θέλουμε τα ταμεία αυτά να είναι υγιή, στιβαρά. Και αν θέλουμε να αποδίδουν, να επιτελούν το έργο τους, πρέπει να παρέχουν εγγύσεις. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα πάμε προς την κατεύθυνση που είπε η Σοφή, να βρούμε με ποιο τρόπο θα είναι πραγματικά ασφαλή τα μία, Γιατί πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι δεν το λαμβάνουμε αυτό υπόψη. Θέλουμε τις εγγύησεις, αλλά δεν θέλουμε να, έχουμε, να λάβουμε το κόστος. Θέλουμε ασφαλείς επενδύσεις. Μα οι ασφαλείς επενδύσεις έχουν τίμημα. Τίποτα δεν είναι τζάμπα στη ζωή. Επομένως, Εάν θέλουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα, θα πρέπει να καταβάλουμε το τίμημα. Έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μία μικρή διαφορά μου είναι ότι μόνο έτσι θα αποδώσουν οι επενδύσεις του πρώτου πυλώνα. Οι συντάξεις του πρώτου πυλώνα, συγγνώμη. Συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Λούντβικ, ότι δηλαδή αν κανείς παρακολουθήσει την προβληματική στο Βέλγιο, το θέμα δεν είναι ότι τα 65 έτη δεν είναι η σωστή ηλικία. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος παίρνει σύνδεξη πολύ πιο νωρί. Μέσω ώρες είναι στο Βέλγιο τα 58. Τα 58. Δεν δουλεύει στο σύστημα. Ας έχει ο κόσμος, επομένως, πλήρη σταδιοδρομία. Και να μην λέμε ότι θεωρητικά παρατείνουμε το, το όριο συνταξιοδότησης. όχι μόνο ο πρώτο πυλώνας, όπως είπε η Σόφη. Αυτά που λέει η Σόφη να εξασφαλίζονται σε όλου του πυλώνε. Ή θα δαπανούμε λιγότερα ή θα υπάρχει μεγαλύτερο εισόδημα για αυτά τα ταμεία, το οποίο αυτό μπορεί να ρυθμιστεί κάπω με, κάποια, με κάποιο είδου ε, έσοδα. Δεν υπάρχει λύση τη ασημένια σφαίρα. Εντάξει. Και εγώ λοιπόν συντάσσω την πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καμάλ. Εδώ έχουμε διάφορες δήματα. Όπως είπε και ο Φιλίπ, ε, πολλές φορές δεν συντάστησα και εγώ σαν τον Φιλίπ με την πλειοψηφία. Αυτή τη φορά συμφωνώ, γιατί πάντως υπάρχουν ε, κάποιοι προβληματισμοί σε σχέση με το τι θέλει να κάνει η Κομισιόν. Πολλές φορές η Κομισιόν θέλει να πανέμβει εκεί που δεν θα έπρεπε, στα εθνικά συστήματα συνταξιοδότησης. Συμφωνώ όμως ότι θα πρέπει να είναι ανθεκτικό το σύστημα, αλλά δεν νομίζω ότι η πολυνομία και η, ρυθμιστική αντιμετώπιση θα φέρει κάτι τέτοιο. Όπως είπαν και οι Θα πρέπει να δούμε πώς τι θα κάνουμε με, με, με την τροπολογία μας. Έχουμε την 112 σε σχέση με <clears throat> κάποιο χρονικό, κάποια προθεσμία. Πώς δηλαδή ο κόσμος θα ενθαρρύνεται να λαμβάνει την ευθύνη της αποζημίωσης. Δεν είπα να είμαστε σκληροί να τους εγκαταλείπουμε, αλλά πρέπει να τους τα πούμε ξεκάθαρα. Το θέμα είναι βέβαια ο καθένας πόσο θέλει να έχει ρόλο δεσποτικό, καταπιεστικό, ρυθμιστικό. Και στη δική μου χώρα υπάρχουν ρηχογνωμίες. Είπα επίσης ότι με κάποιο είδου ε, στάνταρ εναρμόνησης έχω κάποιες ενστάσεις. Επίσης συμφωνώ με αυτά που λέτε για τα ταμεία είναι θέμα αυτό με τη, με τη σύμβαση, τη συνθήκη ε, αξιοπιστία 2. Ότι τα ταμεία μακροπρόθεσμα είναι κάποια επένδυση. Και γι' αυτό και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες. Όχι, δεν έχει λυθεί το βασικό πρόβλημα. Εάν τα πράγματα πάνε στραβά, κάποιος να το κόστος της διάσωσης. Είδαμε τι έγινε με την Lehman Brothers και με την Northern Rock. Ακόμα δεν λύσαμε το πρόβλημα. Τα ταμεία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μακρόπνο. Να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Να εξασφαλίσουμε εκεί ένα περιβάλλον τέτοιο που να, να εμπνέει ασφάλεια με κάποιο τρόπο. Ενία αγορά, όπως λέει η Επιτροπή, αλλά να υπάρχει και η κινητικότητα. Εγώ από τότε που αποφύτησα έχω αλλάξει 6-7 δουλειές και όχι επειδή με διώχνανε, γιατί ήθελα να εξελιχθώ ή να μετακινηθώ από τη μία χώρα στην άλλη. Και θα πρέπει επομένω να δούμε πώς αυτό θα συνδυαστεί η κινητικότητα. Δηλαδή, στην ενιαία αγορά, πώς θα εξασφαλιστεί από τη μια χώρα στην άλλη. Όλα αυτά τα συζητήσουμε με εισηγητή και τους σκιώδες εισηγητές. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον Τόμας Χάντελ. Σιλβί, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Τόμας, για τη δουλειά. Δεν θα προσθέσω και πολλά σε σχέση με αυτά που είπαν οι σκιώδεις, απλώς να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο-τρία σημεία. Πρώτον, όλοι συμφωνούμε για την ενίσχυση της ασφάλειας των συντάξεων, όμως νομίζω ότι το κόστος ε, για τις επιχειρήσεις ε, πρέπει να είναι λογικό και πολλές φορές η λογική φαίνεται πως είναι ε, να βάζουμε στο ίδιο πλαίσιο πράγματα που δεν ανήκουν στο ίδιο πλαίσιο. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και όχι ιδεολόγοι. Λοιπόν, δεύτερον, θεωρώ ότι υπάρχει ε, ένα μεγάλο διακύβευμα στο επίπεδο της κινητικότητας της εργασίας. Δεν πρέπει να το χάσουμε από τα μάτια μας αυτά. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν ε, να δουλέψουν σε μία άλλη χώρα είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το βλέπουμε στην οικονομία, στη θεωρία της οικονομίας και γενικά ειδικότερα της τραγικής κατάστασης στο νότο της Ευρώπης, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο, όμως δεν γίνεται καλή κατανομή των πόρων και γι' αυτό δεν είναι τόσο μεγάλη η συμμετοχή. Πρέπει να το ε, εξετάσουμε αυτό. Τώρα, για την δημιουργία αρχών εποπτείας, ε, ίσως να υπάρχει κάποιος τρόπος να ενισχύσουμε τον έλεγχο των εποπτών, των ελεγκτών και να μην κάνουμε εκ των προτέρων κανόνες. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν σε αυτή την έκθεση και στην ε, αναθεώρηση της ΙΟΠΑ που θα έρθει του χρόνου, αν θα ήταν καλό να έχουμε μια τέτοια ρύθμιση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του καλύτερου ελέγχου για την προστασία των μισθωτών χωρίς να μπούμε τελικά σε ένα ε, νομικό παζλ ε, το οποίο ουσιαστικά θα έχει από τη μία τις ε, ασφαλιστικές εταιρείες και από την άλλη τις επιχειρήσεις ε, που θα προσφέρουν κάποιες, κάποια πλέον εκτήματα. Δεν ξέρω αν είναι εδώ η Κομισιόν, αλλά θα έπρεπε να ακούσει τη φωνή του Κοινοβουλίου, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι αυτό δεν πάει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κυρία Ντόμεν ε, Ρουίτεν. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μπορώ να συνεργαστώ με την Επιτροπή. Έχουμε κοινέ εξουσίες για αυτό το θέμα. Έχω ακούσει πολλά για τις αρμοδιότητες των κοινωνικών υποθέσεων της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα θα πάνε καλά με τον κύριο Μάν. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, κάποιες ε, παρεξηγήσεις που πρέπει να λύσουμε εδώ. Ο πρώτος ε, πυλώνας, μίλησατε για το Ολλανδικό σύστημα και στην Ολλανδία ο πρώτος πυλώνας είναι ο πιο σημαντικός από όλους. Πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Είναι ο πιο σημαντικός και στην Ευρώπη επίσης. Στην ουσία το θέμα είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί ο πρώτος πυλώνας και η ιδέα του Τόμας είναι ότι όταν έχουμε περισσότερους ανθρώπους υγιείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι υπόλοιποι πληρώνουν ασφάλιστα, ασφάλιστρα για τον πρώτο πυλώνα των άλλων. Αν δεν θέλουμε να αυξηθούν τα ασφάλιστρα, θα έχουμε και μικρότερες συντάξεις. Και αυτό είναι κομμάτι της στρατηγικής 2020, ότι όλοι πρέπει να έχουν μια επαρκή σύνταξη. Εμείς λοιπόν στην Επιτροπή Επασχόλησης λέμε ότι ό,τι και αν συμβεί θα πρέπει για κάθε σύστημα, για κάθε πυλώνα να εξοικονομούμε χρήματα έτσι ώστε το βάρος να μην πέσει στους ώμους των επόμενων γενεών. Για το δεύτερο πυλώνα, πρόκειται για ένα σύστημα στο οποίο οι εργαζόμενοι και εργοδότες από κοινού αναλαμβάνουν την ευθύνη να επενδύσουν λίγο περισσότερο από ό,τι δίνεται για τον πρώτο πυλώνα. Στην Ολλανδία έχουμε πολλούς αυτοαπασχολούμενους. Αυτοί πρέπει να πάνε σε έναν τρίτο πυλώνα αν θέλουν περισσότερο εισόδημα. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι ο τρίτος πυλώνας παρέχει και σε επαρκή σύνταξη. Και μετά υπάρχει η συζήτηση σχετικά με τα επιδόματα και τα λοιπά ε, και τις συνεισφορές. Ε, όλο και περισσότερο ο κόσμος πηγαίνει προς ένα σύστημα συγκεκριμένων εισφορών ε, λόγω των διακυμάνσεων στις χρηματιστηριακές αγορές. Πολλές χώρες λοιπόν έχουν κάποια μείγματα μεταξύ των δύο ε, συστημάτων, των ορισμένων επιδομάτων και των ορισμένων εισφορών. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Τώρα, η φορητότητα που αναφέρθηκε. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αν είμαστε ευέλικτοι στην αγορά εργασίας, όταν πηγαίνουμε δηλαδή από την με τον εργοδότη στον άλλον, θα έχουμε εγγύηση για τα συνταξιδοτικά δικαιώματα που έχουμε ήδη σωρεύσει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι ότι το κεφάλαιο που θα έχει κανείς σε ένα συνταξιδοτικό ταμείο θα μπορεί να μεταφέρεται σε ένα άλλο χωρίς καμία δυσκολία. Αυτό βέβαια δεν χρειάζεται εάν τα δικαιώματα που έχεις ε, ήδη κερδίσει είναι εγγυημένα. Όχι μόνο όταν πας ε, στο εξωτερικό, να ισχύει το ίδιο και όταν πηγαίνεις ε, σε έναν άλλο εργοδότη στην ίδια χώρα. Να κάθονται εκεί και να σε περιμένουν τα δικαιώματά σου. Στη Γερμανία Έχουμε μια πενταετή περίοδο. Στα πρώτα πέντε χρόνια πληρώνεις ένα ασφάλιστρο ως ε, ε, εργαζόμενος υπό τον δεύτερο πυλώνα. Αυτό μπορείς να το πας σε ένα συνταξιδοτικό ταμείο άλλο όταν φύγεις. Αλλά το κομμάτι του εργοδότη δεν έρχεται μαζί σου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτό. Μετά από πέντε χρόνια, λοιπόν, να πας σε άλλη, σε, άλλη εταιρεία, δεν έχεις στην ουσία δημιουργήσει επικουρική σύνταξη. Αν λοιπόν ε, ε, τεθεί σε ισχύ αυτό το σύστημα φορητότητας, ίσως θα ήταν καλό να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα ευνοεί αυτή τη μεταφορά των δικαιωμάτων ε, και εντός της ίδιας χώρας και μεταξύ χωρών. Όταν κανείς έχει ε, κατακτήσει συνταξιοδοτικό ε, δικαίωμα, η περίοδος αναμονής θα πρέπει να είναι από 1 έως 5 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί συνάδει και με την κινητικότητα. Για τον τρίτο πυλώνα τώρα, ο κανονισμός που διασφαλίζει ότι τα συνταξιδοτικά δικαιώματα μπορούν να μεταφερθούν από τη μία χώρα σε άλλη. Αυτή τη στιγμή ε, θα πρέπει αυτό που ζητείτε είναι ένα σύστημα πληροφοριών ε, σε κάθε κράτος μέλος, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν πόση σύνταξη θα μπορούν να λάβουν και πώς μπορούν να τη βελτιώσουν. Αυτό το έχουμε στην έκθεσή μας και είναι πολύ σημαντικό. Ένα τελικό σημείο για την ηλιακία συνταξιοδότηση. Σημαντικό είναι, αλλά όχι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή ένας στους τρεις στην Ευρώπη είναι άνω των 55 ετών και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που σας πιέζω, αλλά εδώ σε αυτήν την Επιτροπή πάντοτε με τη δουλειά που έχουμε δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Επειδή είμαι σκιώδης εισηγήτρια για την Φεργιότητα 2 και εφόσον υπάρχει και ο Πίτερ Σκίνερ εδώ, ίσως εγώ ε, γνωρίζω περισσότερα για αυτός από μένα για το θέμα, Ήβα ίσως να γνωρίζει περισσότερα από μένα, αλλά περισσότερα γνωρίζουμε από την Κομισιόν. Είπα ο Πίτερ ότι πρέπει να εφαρμόζεται η φερογγιότητα 2. Να πω ότι δεν είναι ο ίδιος κίνδυνος, γι' αυτό η πλειοψηφία είπε ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται η φερογγιότητα 2. Αυτοί έχουν δίκιο. Γιατί το σύστημα της ε, σύνταξης ε, της απασχόλησης ε, είναι μόνο, δεν είναι διαφοροποιημένο έχει να κάνει... Δεν υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία. Μπορείς να έχεις ε, ποικίλε εταιρείε, ε, ποικίλε ε, εισφορές εργοδοτών ή ασφάλιστρα. Αυτό δεν γίνεται σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Γι' αυτό είναι διαφορετικό και πρέπει να το ε, αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Και δεδομένη της δουλειά που έχουμε κάνει, να πω ότι δεν έχουμε ακόμα επιλύσει το μακροπρόθεσμο πακέτο για την ε, ασφάλεια ζωής στην φερογγιότητα 2 ούτως ή άλλως, οπότε καλό θα είναι να εξετάσουμε τι ακριβώς θα συμβεί στην IROPS όταν την κάνουμε. Το λόγο τώρα στον Τόμας, να είσαι λίγο σύντομος γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Έχουμε μεγάλη συνένεση ότι δεν θέλουμε τη φερεγγιότητα 2, είναι η θέση της πλειοψηφίας. Φυσικά χρειαζόμαστε εξασφαλίσεις και για ε, πτωχεύσεις θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, οπότε ένα σύστημα πληροφοριών που λειτουργεί είναι απαραίτητο. Επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται ε, σε περίπτωση που έχουμε επικουρικές ιδιωτικές συντάξεις, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως θα μπορούσε να μας δώσει λύση εδώ. Επίσης, να πω ξεκάθαρα ότι οι επενδύσεις για αυτές τις ε, ε συντάξεις, τις επικουρικές, έχουν να κάνουν, εξαρτώνται πλήρως από τις αξιολογήσεις των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Έτσι λοιπόν η χρηματοδότηση στο μέλλον δεν είναι δεδομένη και εμείς θέλουμε ασφάλεια. Επίσης, ε, κάποιες σχετικές ε, πληροφορίες με αυτά που είπε ε, η Όλα. Συμφωνώ πλήρως ότι το κομμάτι των νέων είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση και πρέπει να ε, το φέρουμε αυτό στον πυλώνα 2. Δεν πρέπει οι νέοι να τιμωρούνται. Συμφωνώ πλήρως με αυτό που είπες. Φίλιπ, σίγουρα θα δούμε αν είμαστε αρκετά στεναροί. Έχουμε αυτά τα stress tests. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, συντάξεις οι οποίες ε, μπόρεσαν να αντισταθούν στην κρίση και Σιλβί, Θα κοιτάξουμε στην οδηγία Ορπς ε, να δούμε αν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ρύθμιση και επέμβαση. Θα πρέπει ίσως να κάνουμε κάποια, κάποιο συμβιβασμό. Επίσης για την ε, φορητότητα ε, έχω διάφορες θέσεις. Τώρα η συζήτηση δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητα για το 1 έως 5 έτη, για την εισαγωγή στο σύστημα στα 23 έτη κτλ. Τέλος πάντων, χρειαζόμαστε μια κοινή διατύπωση που δεν έχουμε, όμως μπορούμε να βρούμε καλές συμβαστικές λύσεις, ειδικά ε, από κοινού με την Επιτροπή Απασχόλησης, γιατί είναι κοινό μας ε, έργο αυτό, αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. 18 και 19 Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια δεν θέλουμε να το γίνει αυτή η ψηφοφορία και στι στις 21 Φεβρουαρίου θα γίνει η, η, ψήφιση στην Επιτροπή και θα πάμε ε, μετά για την Ολομέλεια του Απριλίου για το θέμα αυτό και τώρα για τη συνέχεια θα δώσω τις σκητάλη στην Αρλίν που αυτή μέχρι την μεσημερινή διακοπή πρόκειται να προεδρεύσει και παρακαλώ επίση οι συνεργάτε των βουλευτών καθόνται στι θέσει του και όχι στι θέσει των βουλευτών. Ελπίζω το ακούσατε όλοι. Οι συνεργάτε, οι βοηθοί στι θέσει των βοηθών. Uh, Από ό,τι βλέπω, ούκαν το πόλο το F όσον αφορά τους παρόντες. Έχουμε τώρα για τα ΟΣΕΚΑ, τους ΟΣΕΚΑ τέλο πάντων, την έκθεση του κυρίου Γιγόλ. Κύριε Γιγόλ μπορείτε να μας παρουσιάσετε το κείμενο ε, έχω αναλάβει και εγώ το θέμα για τους σοσιαλιστές. Γκίγκολτ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ στην αρχή για τις τροπολογίες σας. Αύριο δε θα έχουμε μια συνάντηση ε, με τους ε, σκιώδες και θα ήθελα να έρθουν όσο γίνεται περισσότεροι και έτσι να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά στις λεπτομέρειες τους. Για να δούμε τώρα όλες τις τροπολογίες, να, να δούμε ανά θέμα και επίσης να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες παρατηρήσει να σας πω και εγώ που μπορούμε, πώς να κινηθούμε για κάποιες συμβαστικές. Πρώτα πρώτα επομένως όσον αφορά τις ε, αμοιβέ. Ε, βασικά αυτό που το οποίο θα ήθελα είναι να ευθυγραμμιστούμε με τις ε, αρχές του FSB και επίσης να ευθυγραμμιστούμε με τις θέσεις τις οποίες υιοθετήσαμε όσον αφορά την, την νομοθεσία για την πτώχευση. και με τη θέση που αποκρισταλώσαμε για την οδηγία των κεφαλαιοχικών απαιτήσεων. Θέλουμε να υπάρχει διαχωρισμός για στις αμοιβέ των στελεχών των εταιριών θα πρέπει να κάνουμε μια συμβαστική διάταξη όπου ίσως για τους μικρότερους ΣΕΚΑ και μικρότερες εταιρείε γενικά δεν θα είναι εφικτό αυτό. 62, Μπάλτς, ε, θέλει συνάδελφος, ο Διευθύνων Σύμβουλος να ελέγχει αυτός τα θέματα των αμοιβών. Αυτό όμως θα αντέβαινε στην ε, ε, οδηγία που είπαμε προηγουμένως. Και έχουμε επίσης σχετικά την 61 του Όλε Σμιτ, την 63. Θα πρέπει να δούμε τι θα ακολουθήσουμε. Στο 64 ο κύριος Μαν θέλει να έχουμε ε, μια άλλη αντιστοιχία όσον αφορά τις ε, ε, αμοιβέ και να λάβουμε όμως πάλι υπόψη την οδηγία για τις κεφαλικές απαιτήσει και να είμαστε προσεκτικοί. Στο 65 τώρα, Μπάλτς. Ο κύριος Μπάλτς θέλει οι εθνικές αρμόδιες αρχές να ορίζουν αυτή την ε, αναλογία των αποδοχών. Είπαμε, ε, ε, θα πρέπει να είμαστε εδώ προσεκτικοί γιατί έχουμε την, ήδη έχουμε συμφωνήσει όσον αφορά την επιδιατησία μετά ε, ο κύριο Σμιτ επίση κάτι λέει χρηματοπιστωτικό όμιλο. Προσοχή όμω να μην ε, καταλήξουμε σε μια κατάσταση κατά την οποία να έχουμε ε, αντικίνητρα στην εταιρεία. 68 και 69, Μπάλτς και Σμιτ και οι δύο θέλουν να υπάρχει μια μεταβλητή συνστόση των αποδοχών για τους ΟΣΕΚΑ. Όμως, εδώ υπάρχει συμμετοχή του καταναλωτή και εδώ πρέπει να υπάρχει ψη... μεγάλη ποσότητα καταναλωτή. 67, Σμιτ, διορθώνει κάτι που είναι σωστό. 70, Καμάλ. Και ο Καμάλ θέλει να δει κατά πόσον για τις μικρότερες εταιρείες ίσως δεν θα πρέπει να είναι σωστό να έχουν διαφορετική λειτουργία όσον αφορά τις ε, αποδοχές. Είναι σωστό αυτό και θα πρέπει μένως ε, ε, στις λεπτομέρειες να το, και να το χτενίσουμε και ίσως με καθημερινή γραμμή να δούμε ποια, τι θα όταν λέει, όταν λέει για τις δέουσες αποδοχές, τι θα πει δέουσες για τις κατηγορίες των διαφορετικών εργαζομένων. Προσπαθούμε να βρούμε τώρα μια διατύπωση που να καλύπτει όσο γίνεται περισσότερο σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Έχουμε τις τροπολογίες μας 10 και 20. Έχουμε διαφορετικές προτάσεις, ούτως ώστε να αλλάξει ε, αυτό. Ε, ο Σαΐντ λέει οι εργαζόμενοι. Ε, προσοχή όμως να μην εξαιρέσουμε κάποιους οι οποίοι δεν είναι εργαζόμενοι θεωρητικά, αλλά εργάζονται στην εταιρεία. Άρα να δούμε τις τοπολογίες Μπάλτς και Σμιτ. Και να δούμε μόνο εδώ πέρα να μην ανοίξουμε το παράθυρο σε κάποιο είδου ε, ρυθμιστική επιδιαιτησία. Τώρα όσον αφορά τι υπόλοιπε ε, αποδοχέ επιδόσεων και αποδόσεων, έχουμε εδώ διάφορε τροπολογίε Έχουμε την 122 της Αλήν ε, Μακάρθη ε, σε σχέση με αυτή την ε, βαθμιαία κατάργηση για τους ΟΣΕΚΑ. Επίσης, έχουμε τις τροπολογίες Σμιτ και Μαν που αφορούν το ίδιο ζήτημα. 121 και 123. Θα πρέπει αυτά να ξανασυζητηθούν. Ο κύριος Σμιτ λέει να τα μελετήσουμε καλύτερα. Άρα το θέμα θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, συζητηθεί από τους ε, σχεδόν ηγητές. Έχουμε πολλές τροπολογίες τώρα, Κοζές και Μάν, 72, 73, 75, όσον αφορά κάποιες μεταρρυθμίσεις, τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, 108, 112, 113, επίσης για το ίδιο θέμα και στο τέλος ε, και του Σμιτ υπάρχει μια τροπολογία άλλη, 110, που λέει να μην γίνεται επαναχρησιμοποίηση. Καλά, θα αποσύρω τις δικές μου τροπολογίες και θα προσπαθήσω να κάνω μια συμβαστική τροπολογία με όσα είπαν όλοι. Τώρα όσον αφορά την εκχώρηση κάποιων αποθετικών ε, χρεώσεων ή υποχρεώσεων, depository duties στα αγγλικά. Έχουμε την τροπολογία 76 του Σαΐτ Καμάλ, ο οποίος θέλει την απέτηση του διαχωρισμού να την διαγράψουμε. για τους ίδιους πόρους και τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Δεν ξέρω, μήπως ε, και εδώ πάμε σε κάποιο είδους ρυθμιστική επιδιαιτησία. 77 και 80 του Γκοζές και του Μπάλτς. Συγχαρητήρια γιατί σήμερα έχουμε την 50η επέτειο του Ελιζή συμφωνία του Ελιζέ και βλέπουμε εδώ πέρα πόσο ομονούν Γερμανοί και Γάλλοι. Βλέπετε πώς αποδίδει η συνεργασία. Το δίδυμο αυτό επιτυχία στην Ευρώπη συνεχίζει να λειτουργεί. Αποδοτικά το, το γαλλογερμανικό δίδυμο. Παρακάτω, την 80, θέλουμε εδώ πέρα ε, για τον θεματοφύλακα, συμφωνώ. Στο 78 να μην λέει στοιχεία ενεργητικού και να λέει το μέσα. Και έχουμε και την τροπολογία Λούλινγκ που λέει ότι τα μη ρευστά μέσα. Πώς θα πρέπει να ρυθμιστούν. Καλά να δούμε εδώ πέρα ποια είναι η πιο αρτία δόκιμη διατύπωση. Αλλά να προσέξουμε. Να μην έχουμε αρνητικέ συνέπειε. 72 και 73. Μαν και Γκοζές. για το διαχωρισμό. Να μην υποβαθμιστεί η προστασία του καταναλωτή σε σχέση με τι προβλέπει τώρα το Συμβούλιο. Γι' αυτό και διστάζω να ακολουθήσω αυτό το οποίο υποδεικνύουν. Μετά έχουμε την, τις 84 μέχρι 90, τον Μπάλτς, Γκοζές, Καμάλ, Αν Γένσεν, Όλε Σμιτ και Μαν, διορθώνουν διαφορετικά σημεία του κειμένου. Στο δε της Επιτροπής κάποιε κάποιες ε, εξαιρέσεις όσον αφορά ε, κάποιο δίκαιο τρίτου τρίτης χώρας για το διαχωρισμό, κατά πόσον ε, είναι δυνατόν να αποτελεσματικός ή όχι. Αν κανείς διέγραφε τον διαχωρισμό, τότε δεν θα είχαμε αρκετή προστασία του καταναλωτή. Ούτε θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο είδου ε, επανόρθωση ζημίες. Σύμφωνα με τις προτάσεις Καμάλ, Γκοζές κλπ. Άρα, για να συμβαστώ θα πάω προς την κατεύθυνση των τροπολογιών ή της τροπολογίας Γιάννησεν και Σμιτ. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες ρυθμίσεις για την προστασία έναντι της αφαιρεγγιότητας. Θα πρέπει να δούμε όμως τι, ποιες ρυθμίσεις θα είναι αυτές. Τώρα, τα επιλέξουμε επικα στοιχεία. Καμάλ και Σμιτ. 92, 94, 116, 117, και επ' αυτού θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και θα έχουμε συμβαστική η οποία θα συνάδει με το όσο έχει πει το Συμβουλίο. Για την εποπτεία, για τις κεφαλικές απαιτήσει και σε σχέση με το ρόλο των κοινωνικών τραπεζών που πρότεινε η Αν Γένσεν. Επίσης, Υπάρχει το ε, καυτό ερώτημα του κατά πόσον θα πρέπει να επιτρέπεται η απαλλαγή από την ευθύνη σε περίπτωση που θα υπάρχει κάποιος θεματοφύλακας ή υποθεματοφύλακας σε τρίτη χώρα. Έχουμε εδώ την 103, την παρθμόν 103 τέλο πάντων τροπολογία της Γένσεν, ε, της Λούλιν και άλλων Έχουμε συνομιλήσει με τη βιομηχανία γι' αυτό. Η τάση που διαμορφώνεται είναι ότι πολλοί συνάδελφοι λένε ότι θα πρέπει να χαλαρώσουμε την αυστηρότερη πρόταση της Κομισιόν. Και όλα αυτά όμως είναι αιτίες κινδύνων. έχουμε κάποια κάποια και ενεργητικού που όταν υπάρχουν σε κάποιον υποθεματοφύλακα σε τρίτη χώρα προσοχή να μην είμαστε πιο υπερβολικοί από το Συμβούλιο. Άρα, συμβαστική πρόταση θα μπορούσε να υπάρξει λαμβάνοντας υπόψη την τροπολογία 97 του Καμάλ. Αλλά, σαν προπόθεση να τεθεί, ότι αυτή η εταιρεία διαχείριση θα πρέπει να έχει ασφαλιστεί έναντι του κινδύνου. Του κινδύνου που εγκυμονεί τον έννοιο ο υποθεματοφύλακας σε τρίτη χώρα. Όμως προσοχή να καλύψουμε και κάποιες άλλες χώρες όπου μπορεί να έχει τεθεί προϋπόθεση για μια επένδυση, να, για να γίνει επένδυση, δηλαδή να είναι εκεί ο θεματοφυλακίου παθηματοφύλακας. Προσοχή, ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν μετακυλείται ο κίνδυνος στον καταναλωτή. Τώρα πάμε στις κυρώσεις. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θέλουν κάποιο είδους αυστηρότερη εναρμόνιση το μόνο που κάναμε ήταν να ευθυγραμμίσουμε τη θέση του Συμβουλίου με τη δική μας θέση. Την κοινή θέση MED και MAR. Ότως ώστε να έχουμε ισότιμες συνθήκες συνταγωνισμού. Σχετικά υπάρχει τροπολογία της Μακάρθη και επιφυλάσσουμε για κάποιες τροπολογίες που θέλουν να αλλάξουν αυτή την θέση λέγοντας ότι θα πρέπει αυτά να είναι εθνική αρμοδιότητα. Και θα πρέπει να υπάρχει μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Έχουμε τώρα την τροπολογία 124. Σαν αρχή μιλεί για διοικητικέ κυρώσει που δεν θα πρέπει να αποκλείουν τον υπάρχουν και ποινικέ κυρώσει. Και στο δεύτερο τμήμα ε, αναφέρεται ότι Τόσο δεν, δεν συμφωνώ, γιατί έχουμε και άλλες τροπολογίες. για τις εθνικές αρμοδιότητες. 126 Σμιτ, 127 με βρίσκουν σύμφωνο. Και υπάρχουν και κάποιες προτάσεις, όπως η 128 σε σχέση με την οροφή των κυρώσεων που επιβάλλονται στην θηγατρική. Λίγο για 10% όριο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί έτσι κανείς κάποια εταιρεία θα προστατευόταν από ακόμα πιο αυστηρές κυρώσεις γιατί θα σταματούσε η κύρωση στο 10% της ε, θηγατρικής. Άρα αυτό έχει αρνητικές συνδύσεις. 131 όσον αφορά αυτούς που καταγγέλουν. Και αυτό πρέπει να το φιλομίσουμε τις άλλες θέσεις μας και τώρα όσον αφορά την ετησία έκθεση. Θέλουμε τα θέματα των αποδοχών και εδώ θα πρέπει να ρυθμιστούν με τρόπο διάφανο. να δούμε για να συζητήσουμε την 118. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Το κατά πόσον αυτέ οι πληροφορίε, όπω λέει στην τροπολογία, θα αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο. Όταν υπάρχουν πάρα πολλέ πληροφορίε, δεν, δεν αντέχει ο κόσμο. Τόσο έτσι υπάρχει εδώ πέρα μια παρεξήγηση. 120. Σωστή η τροπολογία με κάρτα. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε να μην έχουμε πάρα πολλές προϋποθέσεις γιατί τελικά δεν θα αποδίδουμε. Τέλος, όσον αφορά αυτούς τους, αυτά τα προστατευτικά όρια για τους καταθέτες, για την ΟΣΕΚΑ και την διαχειριστική εταιρεία, θετικό αυτό που προβλέπετε για, την, για το Ηνωμένο Βασίλειο. 109-111 είναι σχετικές τροπολογίες του Σαΐντ Καμάλ που με βρίσκουν σύμφωνο. Αυτά πρεσβεύω και μετά για τις λεπτομέρειες να τα πούμε με τους ε, σκιώδες. Και τώρα περιμένω να ακούσω τις δικές σας απόψεις για τις τροπολογίες σας και τις τροπολογίες των συναδέλφων. Okay, so, so let's get some... Ευχαριστώ. Α ακούσουμε και κάποιε απαντήσει τώρα από τους σκιώδει εισηγητέ που είναι παρόντες. Όπω είπε Σβέν, θα έχουμε πολλέ ευκαιρίε να μπούμε σε περισσότερε λεπτομέρειε στη συνάντηση των σκιωδών σε αυτό το θέμα. Καταρχά ο Τόμας Μαν από το ΕΛΚ θα απαντήσει. Ευχαριστώ καταρχάς συγχαρητήρια στην έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ. Γενικά φαίνεται ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι θα έχει πλειοψηφία, αλλά στο ΕΛΚΑ έχουμε κάποιε βασικέ παρατηρήσει δεν θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη ρύθμιση που θα ήταν υπερρύθμιση για μας. Επίσης αυτό θα οδηγούσε σε κα... στο κάποιες τροπολογίες από τους Ζαμπόλου, Φόκανεν, Μπάλκ και Σάιρ να υποστηριχθούν από μας. Ίσως αυτό μπορούμε αύριο να το λύσουμε. Να πω επίσης ότι για μας είναι πολύ σημαντική η θέση που έχουμε όσον αφορά τις περιορισμούς ε, για τις μεταβλητές αποδοχές, το κόστος ε, διοίκησης. Επίσης, ε, για την απαγόρευση των τελών που σχετίζονται με επενδύσεις. Επίσης, τα performance fees θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνονται και το θεωρούμε σημαντικό στοιχείο αν ε, κάποιος ε, διαχειριστής ενός ταμείου έχει επιπλέον ε, αποδοχές και δεν υποστηρίζεται τα πόσο ψηλές είναι και από πού προέρχονται, τότε ίσως δεν θα συνάδει αυτό με την αιτήσιο ισολογισμό και έτσι καλό θα ήταν να δούμε σε ποια μορφή δημοσίευσης θα πρέπει να καταφύγουμε. Η απαγόρευση για τα performance fees θα ήταν ένα κίνητρο μεν, αλλά αγνοεί όλα αυτά τα στοιχεία. Ποια είναι, ποιες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των ταμείων. Ε, αυτός που ε, δίνει την εντολή είναι αυτός ε, που θα πληρώνει αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αν θέλουμε πολύ, σημαντικά, πολύ σοβαρά ρυθμιστικά μέτρα, τότε πρέπει να διασφαλίσουμε πρωτοβουλίες ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην περιορίζονται στα ουσοσέκα, αλλά και σε άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα. Ε, τώρα, για τα εναλλακτικά ταμεία επενδύσεων ε, για τις, επιχει... για ε, αποζημιώσεις και τη ρύθμισή τους. Θεωρώ ότι και το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό, όμως αύριο στη συζήτηση θα έχουμε μια εκπροσώπηση όλων των θέσεων. Δεν έχει να κάνει με τον Ζαν Πολ, που του εύχομαι το καλύτερα για αυτά τα 50 χρόνια της Ελιζέ. Ελπίζω ε, να μην ζήσουμε ε, στιγμές σαν αυτές που ζούμε στους δρόμους των Βρυξελών που γλιστράνε παντού, να μπορέσουμε παρά τα χιόνια να πάμε ε, στις ορταστικές εκδηλώσεις για αυτές τις δύο χώρες που αποτελούν έναν καλό κινητήρα που οδηγεί την Ευρώπη. Οπότε Εύχομαι τα καλύτερα για, τη σημαντική, για αυτό το σημαντικό σταθμό στην ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Uh, Ο Γκοζές φυσικά θα μιλήσει για αυτό το θέμα επίσης. Θα μιλήσω ως εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και ως εισηγήτρια από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Νομίζω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά για αυτό το θέμα. Υποστηρίζω πολλές από τις τροπολογίες, ε, καθώς και οι Σοσιαλιστές ε, της Επιτροπής. Ε, και τη γενική του προσέγγιση. Φυσικά δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες ε, για όλα τα θέματα. Οι τροπολογίες μου εμπνέονται από το ότι ε, αυτό είναι τμήμα του πακέτου για τους μικροεπενδυτές που συμπεριλαμβάνει και τα PRIPS. Για μένα η προστασία λοιπόν των καταναλωτών για την ομάδα μου είναι πολύ σημαντική. Υποβάλλω τροπολογίες, ούτως ώστε να εμποδίσουμε τα περιοριστικά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ ε, να χρησιμοποιηθούν ξανά από το θεματοφύλακα. Είναι πολύ σημαντικό μέτρο αυτό για την προστασία των επενδυτών. Η βασική ευθύνη του θεματοφύλακα είναι η διασφάλιση, η διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων. Ε, Επομένω, δεν θα μπορεί ο θεματοφύλακα να χρησιμοποιεί τα χρήματα των ΟΣΕΚΑ για δικό του λογαριασμό. Ε, θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα στην νομοθεσία αυτό το πράγμα. Ε, παρόμοιες τροπολογίες έχουν υποβληθεί από τον κύριο Μαν, από τον Βόρθαν Κλίντς, από τον κύριο Γκοζέ, από την κυρία Γιάνσεν, τον κύριο Σμιτ και θα πρέπει, συμφωνώ, να βρούμε τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό, το ώστε να είναι σωστό το κείμενο, να είναι ξεκάθαρο το κείμενο στη τελική του μορφή. Υπέβαλα τροπολογίες για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη αποκάλυψη πληροφοριακών στοιχείων προς τους επενδυτές. Είναι σημαντικό για το καθεστώς ας πούμε, της ευθύνης να ενημερώνται οι επενδυτές ε, ποιος έχει την ευθύνη ε, για τις ε, πρακτικές δανεισμού του ΟΣΕΚΑ, για τα περιουσιακά στοιχεία που είναι σε κίνδυνο και ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνο για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, όχι μόνο για τα ομόλογα και τις μετοχές. Στις συζητήσει στην ομάδα μου πιστεύουμε ότι πλήρης πληροφόρηση για τις επενδυτικές προοπτικές και ένα κατάλογος όλων των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να δίδονται ε, στους επενδυτές για να αξιολογούν τον κίνδυνο. Είναι μια διάταξη που μπορεί να είναι πολύτιμη και πραγματικά επωφελή γιατί θα ενημερώνει τους επενδυτές για την ύπαρξη των ε, περιουσιακών στοιχείων ε, και για το κόστος της φυλαξής τους σε ό,τι αφορά την αμοιβή για τις επιδόσεις των διευθυντικών στελεχών, φυσικά θα πρέπει τα ισχυρό εισηγητές να το συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Συμφωνώ με, την, με τον εισηγητή ότι θα πρέπει ε, το προσωπικό των ε, ΟΣΕΚΑ να παίρνει τέτοια, τέτοιες αμοιβέ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ε, Τέτοιε συζητήσει κάνουμε σε προηγούμενα νομοθετήματα, στη ΜΥΦΙΤ κτλ και ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το θέμα των, ε, του κόστους και του ωφέλους. Ποιος ε, πληρώνει, επομίζεται το κόστος, ποιος πληρώνει. Ε, είναι πάντα ένα θέμα όταν πρέπει να πληρωθούν επιπλέον ποσά. Ο βασικός μου, το βασικό μου μέλημα είναι να προστατευτεί τελικά ο καταναλωτής και όχι ο κλάδος. Ο κλάδος πιστεύει βεβαίως ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα, αυτές αμοιβέ που συνδέονται με τις επιδόσεις αυτά τα bonus ας πούμε, που συνδέονται ε, με τις, επιδόσεις. Είναι πολύ σημαντικό σημείο, θα πρέπει να το συζητήσουμε, θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες και επίσης συμμερίζουμε την άποψη του εισηγητή ε, που είναι κατά των, της τροπολογίας του ECR για την, το διαχωρισμό των ψηφιακών στοιχείων. Υπάρχει κίνδυνο σε περίπτωση αφαιρεγκαιότητας του θεματοφύλακα ε, τα περιουσιακά στοιχεία ε, τελικά να μην είναι ε, ασφαλή. Θα πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν το διαχωρισμό ή μάλλον θα πρέπει να μειώσουμε τον κίνδυνο. Εγώ και η ομάδα μου θα υποστηρίξουμε αυτές τις τροπολογίες, αλλά θα κοιτάξουμε άλλες τροπολογίες που δεν διαγράφουν το διαχωρισμό, αλλά κοιτάνε κάποιους περιορισμούς. Θα πρέπει όμως να μου αιτιολογήσετε τις ιδέες αυτές πριν φτάσουμε σε συμβασμό, τόσο ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο στόχος των περιουσιακών στοιχείων, ε, ή μάλλον να είναι ασφαλή τα περιουσιακά στοιχεία, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ΟΣΕΚΑ. Αυτές είναι οι προτάσεις μου, όπως συζητήσαμε στην ομάδα εργασίας και περιμένω να δω τι συζητήσεις θα ακολουθήσουν με τους άλλους κοιόδης συζητητές, τόσο ώστε να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Ο Βόλφκαν από τους φιλελεύθερους. Η Άννα Γένσεν είναι η συγγήτρια για τους ε, Άλντε, ε, όμως δεν μπορεί να έρθει. Ευχαριστώ τον Όλε Σμίτ για τις προπολογίες ε, που κατέθεσε, ούτε αυτός είναι εδώ. Εγώ αναφέρω τη σκέψη της συναδέλφου. Μου άφησε ένα χαρτί, το οποίο είναι γραμμένο στα αγγλικά και θα το διαβάσω στα αγγλικά θέλει να επιστήσει την προσοχή ε, στις εξής τροπολογίες ιδιαίτερα. Πρώτα, τις τροπολογίες σχετικά με τους κανόνες αμοιβών. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να πληρώνονται performance fees στην ε, εταιρεία διαχείρισης. Το βασικό στοιχείο της ρύθμισης αυτών των αμοιβών είναι ότι οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εταιρείας και ε, προσωπικού. Επειδή το ΙΟΣΕΚΑ ε, πληρώνει performance fees ε, στην εταιρεία διαχείρισης, δεν σημαίνει ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, γιατί και οι δύο θέλουν καλύτερες αποδόσεις. Έτσι λοιπόν, μπορεί αν δεν, υπάρχει, αν δεν υπάρχουν αυτές οι αμοιβέ να μην... Να λαμβάνεται υπερβολικός κίνδυνος. Να λαμβάνεται κίνδυνος. κατά συνέπεια οι επενδύσεις ε, δεν θα ε, πρέπει να ε, ξεπερνούν σε κίνδυνο αυτά που ορίζεται στην οδηγία ως ΕΚΑ. Για την τροπολογία 33 του κυρίου Καμάλ, την 57 και την 58 και την 59 του Σμιτ λέει ότι αναφέρεται η ηγεσία, οι διαχειριστές κινδύνου που λαμβάνουν αμοιβέ θα πρέπει να ε, διαγραφούν, θα πρέπει οι κανόνες ε, να είναι συγκρίσιμοι σε όλους τους τομείς ε, του χρηματοπιστωτικού τομέα και οι συγκεκριμένοι κανόνες δεν είναι σε αυτά τα πλαίσια. Για την 61 και 62 Σμιτ και Μπάλς οι τροπολογίες προτείνουν αλλαγές που είναι παρόμοιες με μία διάταξη ε, στην ε, πρόταση για την ε, οδηγία για τις κεφαλαίκες απαιτήσει. Θα πρέπει λοιπόν να είναι συγκρίσιμες οι διατάξεις. Για την 66 του Μπάλτ στην πρόταση για ένα νέο άρθρο 14, προτείνεται οι εταιρείε διαχείρισης να πρέπει να αποκαλύπτουν συνολικά και σε πληροφορίες ε, για τις αμοιβέ. Δεν λέγεται ακριβώς τι είναι αυτό. Θα πρέπει να έχουμε έναν κατάλληλο ορισμό, γιατί είναι 65 του Μπάλς, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι απαραίτητο να, η μία αρχή να θέσει ε, ε, την αναλογία μεταξύ των μεταβλητών και συγκεκριμένων αποδοχών. Αυτά πρέπει να είναι ισορροπημένα. Το σταθερό κομμάτι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της συνολικής αμοιβή έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία για τις μεταβλητές αποδοχές όπως ε, και τη δυνατότητα να μην δίνονται μεταβλητές αποδοχές. Αυτό είναι πολύ σημαντική διάταξη. Αν ε, η αρχή ε, θέσει αυτή την αναλογία, δεν θα υπάρχει ευελιξία για τις εταιρείε τελικά. Τέλος, ε, για το καθεστώς ευθύνης θα ήθελα να ξέρω γιατί η Επιτροπή αποφάσισε να έχει ακόμα πιο αυστηρές διατάξεις ε, για τους θεματοφύλακες έκα από ό,τι είχαμε στο IFND. Συγκεκριμένα σε επίπεδο υποθεματοφυλακής. Αν δίνονται χρηματοπιστωτικά μέσα σε τρίτο μέρος, τότε ο θεματοφύλακας είναι υπεύθυνο για την απώλεια. Θεωρώ ότι η ευθύνη του θεματοφύλακα είναι δυσανάλογη με τις αντικειμενικές του δυνατότητες. Αυτά. Ελπίζω να είναι εδώ αύριο και να είναι και στη συνάντηση που αναφέρατε. Να πω στο τέλος ε, δύο πράγματα δικά μου. Εγώ ε, κατέθεσα πολύ λίγες τροπολογίες, απλώς ήθελα να πω ότι θεωρώ στην ουσία σημαντικό η ε, οδηγία ο ΕΚΑ ε, να μιλά για τον περιορισμό, τον περιορισμό της περαιτέρω χρήσης ε, των ε, επενδυτικών ταμείων που αφορούν στα AIFM. Το είπαν όλοι οι προηγούμενοι στο ΣΕΚΑ θα πρέπει, στους ΣΕΚΑ θα πρέπει να εξετάζουμε την ασφάλεια των επενδυτών, ειδικά όταν πρόκειται για μικροεπενδυτές. Όσον αφορά τώρα στα χρήματα, στις διοικητικές ε, δαπάνες, ε, δεν υπάρχει κάποια ποσοτικοποίηση. Ε, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς γιατί πρέπει να έχουμε κάποιο περιθώριο δράσεως κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ. Ε, Mr. Kamal, on behalf of the ECR. ECR, Kamal. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς τον συζητητή που μας επέτρεψε την περασμένη εβδομάδα σε τριμερή διάλογο να συζητήσουμε και να διευκρινίσουμε κάποιες από τις τροπολογίες. Τρία βασικά θέματα για τις αμοιβέ. Υπέβαλα τροπολογίε, με σκοπό να διευκρινίσουμε ότι η πολιτική αμοιβών ε, μειώνει τον κίνδυνο και λαμβάνει υπόψη όλα τα συμφέροντα. Ε, πρέπει να δούμε τι κίνδυνοι υπάρχουν, ε, γιατί ως ΕΚΑ επενδύουν για λογαριασμό των επενδυτών. Πριν από λίγα χρόνια, ε, όταν συζητούσαμε την ε, τρίτη οδηγία της κεφαλαιοκές απαιτήσει, συζητούσαμε αυτό το θέμα των αμοιβών. Το θέμα είναι, είναι κατάλληλο να εφαρμόσουμε κανόνες αμοιβών σε άτομα ή οντότητες ε, όταν υπάρχει κίνδυνος για τον ισολογισμό. Για... Συμφωνώ με τον Βόλφ για τον θεματοφύλακα. Καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν δεν θέλει ή μάλλον εξετάζει την ευθύνη του θεματοφύλακα. Ε, με τις τροπολογίες μου προσπαθώ να λάβω υπόψη με την κατάσταση όπου ένα ταμείο, ένας οργανισμός θέλει να επενδύσει σε μια συγκεκριμένη χώρα για να αποφύγει ε, οποιαδήποτε παράπονα ας υπο, ας, ε, από μια φανταστική χώρα, ας πούμε. Και ο θεματοφύλακας λέει, ε, ε εγώ δεν θεωρώ ότι είναι προβληματική χώρα, επενδύω. Ε, επενδυ, επιμένει ο διαχειριστής δηλαδή του ταμείου θα το επιτρέψουμε. Ποιο θα έχει την ευθύνη. Ε, ο θεματοφύλακα δεν θέλει να λάβει την ευθύνη και θα οδηγηθούμε σε διάξοδο. Εμεί λέμε αυτή τη στιγμή α, ο θεματοφύλακα να έχει οπωσδήποτε την ευθύνη. Εγώ λέω να υπάρχει μια συμβατική απαλλαγή ε, στο βαθμό που συμφωνούν και τα δύο μέρη ότι ο διαχειριστή θέλει να επενδύσει αυτή τη χώρα. Τότε η... απαλλάσσεται από την ευθύνη. Κάποιο όμω μου είπε σήμερα ότι τελικά την ευθύνη κάποιο πρέπει να την αναλάβει. Δεν θέλω οι επενδυτέ να αρχίσουν να ταξιδεύουν ανά τον κόσμο για να δουν ποιο θα μηνύσουν σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να είναι είτε ο διαχειριστή είτε ο θεματοφύλακα που θα είναι υπεύθυνο. Και όταν υπάρχει διαφωνία, ίσω ε, αν ας πούμε, ο διαχειριστή πιστεύει ότι είναι αρκετά ασφαλέ, τότε μπορεί να μεταφέρει την ευθύνη του, α πούμε, στο θεματοφύλακα. Δεν είναι η ιστορία μα και η πρόθεσή μα δεν είναι να πούμε στου επενδυτέ, άντε, πηγαίνετε ένα ταξιδάκι για να δείτε ποιο είναι υπεύθυνο. Αν ο διαχειριστή δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί έχει την ευθύνη ο θεματοφύλακα, θα πρέπει να δούμε μήπω έχει την ευθύνη αυτή. Αυτός. Εγώ θέλω να γίνει επίσης ε, λειτουργικός διαχωρισμός και όχι νομικός διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων. Ε, αυτά για τους θεματοφύλακες. Ε, για τις αμοιβέ για τις επιδόσεις. Συμφωνώ με κάποιους από τους συναδέλφους. Ε, γιατί να πληρώνται κάποιοι τόσο καλά και παχυλά όταν ας πούμε δεν τα έχουν πάει τόσο καλά τα ταμεία τους. Συμφωνώ με τον κύριο Μάντερ ότι υπάρχουν τομείς όπου όταν τα πάει καλά ο οργανισμός στο ταμείο ΣΕΚΑ, ας πούμε, τότε να τους αμείβουμε για αυτόν τον λόγο. Αλλά υπάρχει μια πολιτική δυσκολία και διαφωνία μεταξύ μας. Ε, δεν ξέρω, πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό ή να το αφήσουμε για επόμενη διαπραγμάτευση των ΟΣΕΚΑ. Υπάρχουν κάποια, κάποιες αμοιβέ, κάποια μπόνους ας πούμε που μπορούμε να εντοπίσουμε, που μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και κάποια άλλα να τα ξεχάσουμε. Ούτως ώστε να αμείβουμε και να ανταμείβουμε κάποιους όταν τα πηγαίνουν καλά και όχι ό,τι και να κάνουν ας πούμε, καλά κακά. Φυσικά τι εννοείται επίδοση έχει σημασία εδώ. Σε ποιο πλαίσιο τον ορίζεται. Και υπάρχει και μια σύγκρουση συμφερόντων. Και εδώ θέλουμε να το ρυθμίσουμε αυτό το θέμα τη σύγκρουση συμφερόντων, λέει η Πρόεδρο. Ο κ. Γκοζέ θέλει να πάρει το λόγο. Δεν υπάρχει κανένα από την ΚΟΕ. Οπότε α δώσω το λόγο στον κ. Γκοζέ. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σα φάω πολύ χρόνο. Από τις 9 το πρωί είμαι εδώ και ακούω πάντω γιατί δεν είμαι εισηγητή, ακούω απλώ. Το μόνο που θέλω να τονίσω είναι το εξή. Ο εισηγητή έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Το θέμα είναι, που θέλω να σταθώ, είναι το θέμα τη ευθύνη. Σε όλα τα κείμενα που είδαμε, ακόμα και για του οίκου αξιολόγηση, οι επαγγελματίε προσπαθούν ούτω ώστε να έχουν τη λιγότερη δυνατή ευθύνη. Εγώ δεν είμαι κατά των ε, εργαζομένων στον κλάδο το χρηματοπιστωτικό, αλλά νομίζω ότι αυτό το θέμα τη ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλη η υπόλοιπη νομοθεσία δεν έχει κανένα νόημα εάν δεν έχουμε κανόνε για την ευθύνη που είναι ξεκάθαρη. Σε ό,τι αφορά το θεματοφύλακα, οι κανόνε πρέπει να είναι ξεκάθαροι. Γιατί ποιο είναι ο θεματοφύλακα, αυτό που ε, εγγυάται την αποκατάσταση και επιστροφή των κινητών αξιών και των άλλων στοιχείων στους νόμιμους δικαιούχους. Και δεν θα πρέπει εδώ πέρα να αφαιθούμε σε ιδέες ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας διακαονισμός, θα πρέπει να τον απαλλάξουμε κτλ. Πάνω από 25 χρόνια ήμουν δικηγόρος και ξέρω πολύ καλά ότι γύρω από αυτά τα θέματα γίνονται άπειρες δίκες. Λοιπόν, αυτός που ε, διαχειρίζεται την όλη επιχείρηση ε, είναι υπεύθυνος. Ε, εάν, ας πούμε, ο θεματοφύλακας όταν προσλαμβάνει ένα υποθεματοφύλακα, έτσι επειδή θέλει, ας πούμε, τότε παρόλα αυτά κρατάει την ευθύνη. Ε, βέβαια, είναι διαφορετικά τα πράγματα αν το επιβάλλει η εθνική νομοθεσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα, ας πούμε, κάποιων χωρών κτλ. Θυμάμαι τις μεγάλες συζητήσεις που κάναμε ε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το θέμα της ευθύνη. Τα πράγματα είναι απλά. Αν θέλει κάποιο να δώσει απαλλαγή από την ευθύνη, ας το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Αλλά προσοχή, ε, τη στιγμή την κρίσιμη θα πούμε ότι δεν ήταν σαφή τα θέματα της απαλλαγής, ε, όλα τα θέματα μπλεγμένα. Επίσης, για την ασφάλεια. Οι ασφάλειες ασφαλίζουν τους κινδύνους, τους γνωστούς, τους απτούς. Αλλά οι μείζονες κίνδυνοι του να έχουμε έναν ε, θεματοφύλακα σε μία μη ασφαλή χώρα Υπάρχουν προβλήματα με το δίκαιο για την πτώχευση. Ποτέ ένας σοβαρός δικηγόρος δεν θα σας διαβεβαιώσει ότι ο κίνδυνος είναι ξεκάθαρος. Υπάρχει κίνδυνος, δεν υπάρχει κίνδυνος. Πάντα θα υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις. Επομένως, για την ευθύνη δεν πρέπει να είμαστε μαλθακοί. Δεν πρέπει να δώσουμε ευθύνη σε κάποιον αν δεν χειρίζεται τα γεγονότα. Αλλά να μην μπούμε και σε μια κατάσταση όπου θα αφήνουμε όλα στην τύχη και ποτέ δεν θα πούμε κάτι το οριστικό. Όλες οι ασφάλειες θα βάλουν, ας πούμε, στα μικρά γράμματα ε, κάποιες ε, προϋποθέσεις που τελικά θα καταστήσουν την ασφάλεια μη αποτελεσματική. Πολύ ε, σόφρονα όλα αυτά που είπε ο κύριος Γκοζές, θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στη συνάντηση των σκιωδών. Σφέν. Οι διερμηνείς μου δίνουν 5 λεφτά έξτρα. Θέλεις 5 λεφτά ακόμα. Γιατί τελείωσε ο χρόνος. Θα είμαι πολύ σύντομος. Όχι, θα δώσω καλύτερα 2 λεφτά στην Κομισιόν και 3 σε σένα. Η Κομισιόν θέλει να μιλήσει. Uh, okay, but um, I'm going to give you two minutes and I'm going to put it on the clock. If that's okay. Uh, thanks a lot. Uh, δύο και μετά τρία. Ευχαριστούμε. είναι ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού που διαχειρίζεται κάποιος. Από εκεί καθορίζεται το performance fee. Για την επαναχρησιμοποίηση δεν είπαμε τίποτα. Γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει επαναχρησιμοποίηση των στοιχείων αυτών του ενεργητικού. Και είναι πάρα πολύ κακό να λέμε ότι ο διαχειριστής μπορεί να δώσει έγκριση για τέτοια που να χρησιμοποιήσει, γιατί τότε θα παίζει με τα στοιχεία του ενεργητικού ο θεματοφύλακας. Για την πτώχευση τώρα υπάρχει ίση μεταχείριση. Είτε είναι ο θεματοφύλακας σε τρίτη χώρα, είτε είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν έχουμε πτώγευση του υποθεματοφύλακα, θέλουμε η περιουσία της ε, εταιρεία που την οποία φυλάσει να είναι ασφαλής. Και εδώ η συμμεταχείριση, είτε είναι τρίτη χώρα, είτε είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα η συμβατική απαλλαγή, το καυτό θέμα, δεν, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο για τον ΟΣΕΚΑ, αλλά για τον μικροπενδυτή αυτός πώς να ξέρει ποιο να μείνει σε τρίτη χώρα. Ακόμα και αν υπάρξει απαλλαγή πάντως, πάλι κανείς μπορεί να υποβάλει μήνυση. Μπορεί όμως να λυθεί το θέμα μέσω ασφάλισης. Δεν το είπαμε όμως γιατί ακόμα και υπάρχει ασφάλιση πάλι θα πρέπει να προηγηθεί μήνυση. Αλλά πάντως έτσι και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα για τον μικροπενδυτή αν μιλάμε για τρίτη χώρα. Ευχαριστούμε που ήταν τόσο. Και απαντήστε το που με προβληματίζει. και θυμάμαι ότι είχαμε δουλέψει ε, στην, στην, νομική επιτροπή και είχαμε πει ότι πόσα ενοχικά δίκαια πόσων χωρών πρέπει να συντρέχουν. Δεν έχει πάρα πολύ δουλειά να ακούσουν. Πάντως όσον αφορά τα performance fees, η θεωρία ότι θα εξαρτάται 100% η απόδοση και θα συνδέεται με το συμφέρον του επενδυτή, ωραίο είναι θεωρητικά. Πρακτικά όμως είναι δύσκολο να συνδεθεί το ένα με το άλλο και έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτε στην αγορά. Λένε ότι έτσι δεν έχουμε τόσο πολύ ευθυγράμμιση όσο κατάχρηση του συστήματος. Και ευχαριστώ την Κομισιόν που το επεσήμανε. Δεν χρειάζεται να γίνει τέτοια σύνδεση. Γιατί αν υπάρχει ένα ταμείο το οποίο αποδίδει καλά θα έχει για, του για τους ΟΣΕΚΑ έτσι και καλέ επιδόσεις και αναλογικά προράτε επομένω θα αμείβει. Ακριβώς αυτό που είπε και ο Σαΐντ. Και φυσικά και ο μάνατζερ που δουλεύει καλύτερα πρέπει να αμείβει και περισσότερο. Για να δούμε τώρα, τα, τα, τα, τα, πιο τεχνοκρατικά. Υπάρχουν θέματα πολλά με το performance fee και άρα το κοινοβούλιο πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το άλλο θέμα το οποίο ετέθη και συμφωνήσαμε είναι η επαναχρησιμοποίηση. Συμφωνήσαμε. Άλλο. Ευθύνη. Ευχαριστώ τον Ζων Πολ Γκοζές. Όπως πάντα σχεδόν συμφωνώ και επί του προκειμένου. Πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί για αυτό το θέμα. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε εδώ είναι ότι το κείμενο LFMD βέβαια είναι διαφορετικό σε σχέση με το AIFM. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία ταμείων που αφορά τους μικροεπενδυτές. Έτσι κι αλλιώς εμπλέκονται με τους ΟΣΕΚΑ, αλλά θα πρέπει όπως και να είναι να αισθάνονται ασφαλείς. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να ρυθμίσουμε, μην θεωρούμε ότι είναι τα Άγια των Αγίων και δεν μπορώ το αλλάξουμε. Προσοχή και με την επικάλυψη. Συμφωνώ πάντως για την ευθύνη η Επιτροπή ότι δεν είναι δυνατόν να, να αντιγράψουμε το όσο προβλέπει το ένα κείμενο στο άλλο. Πρόεδρε, ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και του διερμηνεί που κάθισαν λίγο παραπάνω για να μπορέσουμε να τελειώσουμε για αυτέ τι προτάσει. Οπότε τώρα θα δούμε τι θα πούμε με τους ε, σκιοδησίτες. Άρα στις 3 η ώρα αρχίζει η ψηφορία για όσους δεν ήταν. Θα τα πούμε αργότερα.